Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλοχαιρετίζω θερμά όλους σας. Με κάποια μικρή καθυστέρηση. Έχω όμως την εντύπωση ότι όλοι δυσκολευόμαστε σήμερα να φτάσουμε στις Βρυξέλλες, διότι οι γεωργοί με τα τρακτέρ τους είναι καθοδόν. Σας καλωσορίζω λοιπόν και σας καλοχαιρετίζω. Ανακοινώσεις δεν έχω τίποτα καινούριο να σας εκθέσω. Πιθανότατα αύριο θα έχουμε κάποιες πληροφορίες, διότι θα έχουμε απόψε συνάντηση συντονιστών. Χαιρετίζω θερμά τον Γενικό Γραμματέα για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριο Χωσέ Μανουέλ Σίλβα Ροντρίγεθ. Ελπίζω να πρόφερα κάπως σωστά το όνομά σας. Σας χαιρετίζω θερμά, σας ευχαριστώ που είσαστε παρόν εδώ. Θέλουμε να δραχθούμε τις ευκαιρίες μαζί σας να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και ελπίζουμε από εσά να έχουμε την έκθεση που θα μας εκθέσετε για την παρακολούθηση. Έχετε τον λόγο κύριε Γενική Γραμματέα. Ξεκινήστε και μετά θα υπάρχει η ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις οι συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε. Έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε Ρόιλ, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου προσφέρετε αυτό το απόγευμα να σας παρουσιάσω τη δεύτερη έκθεση για την παρακολούθηση του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα του 2008. Καθώς είναι η πρώτη φορά που έχω αυτή την τιμή να σας συναντήσω σε αυτή τη νέα κοινοβουλευτική θητεία, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ όσους δεν έχω συγχαρεί προσωπικά και επιπλέον πιστεύω ότι ανεξάρτητα από το κάνοντας λόγο για την έκθεση για το monitoring πιστεύω ότι θα μπορούσαν και άλλα θέματα να καλυφθούν από τα οποία έχω επιλέξει τρία αλλά είμαι στη διάθεσή σας και είμαι πρόθυμος λογικά στη συζήτηση μαζί σας να καλύψω οποιοδήποτε θέμα θεωρείτε εσείς ε, ότι είναι σκόπιμο τα τρία θέματα που είναι σημαντικά νομίζω είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 7ου προγράμματος πλαισίου, η απλούστευση, και τα Joint Technology Initiatives, κοινέ πρωτοβουλίες ε, για την τεχνολογία, για την έρευνα. Καθώς πολύ καλά γνωρίζετε, ιδιαίτερα τα μέλη, τα οποία είναι παλαιότερα μέλη στην Επιτροπή Ήτρε, ο Επίτροπος Ποτόσνικ παρουσίασε στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο αυτής της, πρώτης, αυτής της χρονιάς, την πρώτη έκθεση για την παρακολούθηση, monitoring για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Σήμερα είμαι εγώ εκείνος που θα σας παρουσιάσει τη συνέχεια. Το επόμενο. Τώρα δεν έχω την πρόθεση από πλευράς μου να κάνω μια εξαντλητική παρουσίαση. Αλλά απλά θα επικεντρωθώ στα θέματα εκείνα, τα οποία θεωρώ ότι είναι και τα πιο σημαντικά. Η έκθεση αυτή βασίζεται σε ένα σύνολο δικτών δικτών indicators που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων που συσχετίζονται με την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να αναφέρει κανείς εκείνα που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των όσων συμμετέχουν, την ποιότητα των διαδικασιών αξιολόγησης και την χρήση των νέων μέσων εργαλείων του προγράμματος. Το νέο σύστημα monitoring είναι επίσης ένα από τα κυριότερα εργαλεία της νέας στρατηγικής για την αξιολόγηση των προγραμμάτων πλαισίου. Χάρη στην συστηματική χρήση αυτών των δικτών κατά τη διάρκεια των ετών μπορεί να γίνει μια ανάλυση, ας το πω έτσι, κάθετη για την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Και έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρξει μια πραγματική, αυθεντική αποτίμηση, πιστεύω. Πρέπει επίση να προσθέσω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό μέσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων πλαισίου. Η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια εξαντλητική αποτίμηση αξιολόγηση των προγραμμάτων πλαισίου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία που είναι θεμελιωδου σημασια για αυτά. Θα ξεκινήσω με τι ε, προκηρύξεις ε, για την υποβολή προτάσεων. Κατά τη διάρκεια των δύο ε, πρώτων ετών Ζωή αυτών των προγραμμάτων 25.000 αιτήματα διατυπώθηκαν με περίπου 150.000 συμμετέχοντε, που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά αυτά τα νούμερα, αυτοί οι αριθμοί. Και από αυτούς 5.500 δηλαδή εγκρίθηκαν με μια συνολική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Α, έτσι επωφελήθηκαν συνολικά 33.000 συμμετέχοντες. Και αυτό είναι κάτι παραπάνω από το 20% όσον αφορά τους συμμετέχοντες που είχαν θέσει αιτήματα. Πέρα από αυτή τη σύντομη αναδρομή στην ιστορία, για πρώτη φορά οι προκηρύξεις για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ξεκίνησαν μία εβδομάδα πριν από την έναρξη σε ισχύ του πρόγραμματος πλαισίου. 22 Δεκεμβρίου δηλαδή του 2006 όταν αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτά είναι προφανή στοιχεία για μας σήμερα πια και αποτελούν τμήμα του κανονικού κεκτημένου. Είναι πράγματα που ποτέ δεν θα μπορούσαν να είχαν δρομολογηθεί και να έχουν υλοποιηθεί σε προηγούμενα προγράμματα πλαίσια. Καθώς γνωρίζετε, είναι ανοιχτά σε όλους αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο, στα πανεπιστήμια, κέντρα έρευνας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις δημόσιες διοικήσεις και αρχές καθώς επίσης και κοινοτικές αρχές και θεσμικά όργανα, καθώς επίσης και ιδιώτες συμμετέχουν σε, αυτά τα, σε αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο. Τα πιο συχνά, το, οι πιο συχνή είναι τα κέντρα διδασκαλίας και πανεπιστημιακά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ, που καθώς γνωρίζετε αποτελούν μεγάλο μήμα σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή με το 15,5% των εποφελουμένων κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών του προγράμματος πλαισίου. Πάνω από δύο τρίτα αυτών των ΜΜΕ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμμετέχουν στο πλαίσιο συνεργασίας και πάνω από ένα τέταρτο από αυτές στο πρόγραμμα των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που καθώς ξέρετε έχετε, έχει ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο τμήμα που στοχεύει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνεχίζοντας κάπως τα στοιχεία για τη συμμετοχή και εξετάζοντας τη διεθνή συμμετοχή θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχουμε το πρόγραμμα έρευνας που είναι το πιο διεθνές στον χαρακτήρα του από όσα υπάρχουν σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα. 136 χώρες 136 χώρες εκπροσωπούνται στις δραστηριότητες του προγράμματος πλαισίου. Ανάμεσα μεταξύ αυτών των τρίτων χωρών που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι η Ρωσία, η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική ισότητα, που και αυτό είναι ένα πολιτικό, πολύ σημαντικό θέμα για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, το 21% των ερευνητών, κύριων ερευνητών ή αρχηγών επικεφαλής ομάδων ήταν γυναίκες. Και αυτό το ποσοστό ανεβαίνει σε πάνω από 35% στις δράσεις, δράσεις Marie Curie. Καθώς γνωρίζετε, αλλά η πολίτητα για την ισότητα αποτελεί μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας διασφαλίζω ότι θα συνεχίσουμε την παρακολούθηση και εξέλιξη αυτών των δικτών πάρα πολύ προσεκτικά εκ του σύνεγγης. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σας ενημερώσω και για ένα στοιχείο θεμελιώδες για αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο που είναι το σύστημα αποτίμησης, αξιολόγησης, που είναι ένας από τους πυλώνες, τους άξονες του συστήματος. Σε μία από τις παλαιότερες προηγούμενες παρεμβάσεις μου στην ίδια αυτήν κοινοβουλευτική επιτροπή είχα αναφέρει τη σημασία που δίναμε στην αξιολόγηση και την ανεξαρτησία που πρέπει να χαίρει το σύστημα αξιολόγησης. Και έτσι ποτέ δεν θα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αλλαγή των ε, θεμάτων. Δεν έγινε αυτό τα δύο χρόνια που ισχύει αυτό το πρόγραμμα, ούτε έχω υπόψη μου να ζητήσω κάποια τέτοια αλλαγή, ανατροπή στα επόμενα δύο χρόνια που απομένουν. Η ποιότητα λοιπόν της αξιολόγησης ήταν θεματοποιήθηκε ως ικανοποιητική ή εξαιρετική βαθμολογήθηκε για το 98% των, των ε, ε, όσων συμμετείχαν στην αξιολόγηση και όσων συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογών κατά τη διάρκεια του 2008. Όμως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι το 96% αυτών των αξιολογητών θεωρούν ότι οι δικές μας διαδικασίες αξιολόγησης είναι ίσες ή ακόμα και καλύτερες από εκείνες που υπάρχουν στις υπόλοιπες χώρες ή στον υπόλοιπο κόσμο και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να το θεωρήσουμε σαν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, σαν ένα σημαντικό, ας το πω έτσι, εμβληματικού χαρακτήρα στοιχείο του 7ου προγράμματος πλαισίου. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι η διαδικασία επιλογής μας να μπορεί να έχει αυτές τις πάρα πολύ υψηλές προδιαγραφές για την ποιότητα. Αυτές οι υψηλές προδιαγραφές για την ποιότητα επίσης επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα όσον αφορά τις, ε, τα αιτήματα για τη ε, διαδικασία αξιολόγησης. Καθώς γνωρίζετε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έχουμε εισαγάγει μια διαδικασία της ε, αμφισβήτησης ή ας το πω έτσι ε, εξέτασης της ε, αξιολόγησης, redress procedure, 25.000 από τις περίπου 25.000 αξιολογήσεις, 1.170 υπήρξαν αντικείμενο κάποιας προσφυγής, αλλά μόνο 17 οδήγησαν σε μια αναθεώρηση της αξιολόγησης, οδηγήθηκαν σε αναθεώρηση, πράγμα που είναι, ας το πω έτσι, αμεληταία ποσότητα. Και πιστεύω ότι και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει όλους να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Τώρα τέλος, εν τέλει, όσον αφορά την διαδικασία απλούστευσης, θα ήθελα να σας πω το εξής. Είχαμε μεγάλη βοήθεια που δόθηκε στα, με τα σημεία των εθνικών συνδέσμων, εθνικών ε, σημείων επαφής και επιβεβαιώθηκαν οι πρόοδοι το στη διαδικασία απλούστευσης στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιος πλαίσιο σε σχέση πάντα με τη σύγκριση με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. 70% των περιπτώσεων θεωρείται ότι στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο έχουμε ε, προκηρύξεις, ε, έντυπα και διαδικασίες που είναι καλές ή εξαιρετικές και πιο απλές σε σχέση με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Οπωσδήποτε αυτό που θα ήθελα να σας πω και θα το δούμε αυτό μετά, αυτό το επίπεδο ικανοποίησης για μένα προσωπικά είναι κάτι που δεν με κάνει να είμαι ικανοποιημένος και σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα και θα σας δώσω κάποια στοιχεία σχετικά με αυτό το θέμα και την προσωπική μου βέβαια δέσμευση να συνεχίσουμε την πορεία προς βελτιώσεις σε αυτή τη διαδικασία στο μέλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά ήταν τα θεμελιώδους σημασία στοιχεία για το monitoring, την παρακολούθηση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Και λογικό είναι ότι και οι υπηρεσίε μου και εγώ είμαστε απόλυτα πρόθυμοι και στη διάθεσή σας, ώστε γραπτώς ή προφορικά να σας δώσουμε οποιαδήποτε στοιχεία επιθυμείτε για αυτά τα αριθμητικά μεγέθη που προαναφέρθηκαν. Θα ήθελα τώρα τη σειρά μου να αναφερθώ σε κάθε ένα από αυτά τα τρία πρόσθετα θέματα που θα ήθελα να σχολιάσω μαζί σας. Το πρώτο από αυτά είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά τη διάρκεια του 2009 η Γενική ε, Διεύθυνση για την Έρευνα προβλέπει όπως ε, κάθε χρονιά και ήταν αυτό η ρήτρα κάθε έτος μία τέλεια εκτέλεση των κονδυλίων του προπολογισμού και σε πιστώσει υποχρεώσεων και σε πιστώσει πληρωμών. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέχρι σήμερα, το ποσοστό εκτέλεση ε, του έτου είναι 86 περίπου σε πιστώσει υποχρεώσεων και 56% <clears throat> περίπου σε πιστώσεις, 57% ε, με συγχωρείτε, σε πιστώσεις πληρωμών και περίπου 2,3 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια ενώ συνόλου 4 δις ευρώ πληρώθηκαν στους ε, ε, όσους εμπλέκονται και εποφελούνται. Αυτά τα στοιχεία στη σημερινή ημερομηνία είναι συγκρίσιμα και παρόμοια με τα προηγούμενα έτη συγκρίνοντας αυτή τη στιγμή. Αλλά να πάρουμε το 2008 για παράδειγμα. Κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου, γύρω στις 7 το βράδυ, ο Γενικός Διευθυντής για τους Πόρους απευθύνει ένα SMS και με ενημερώνει για το ποιο ήταν το επίπεδο εκτέλεσης. Το επίπεδο εκτέλεσης του 2008 ήταν 99,89% σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 99,85% σε πιστώσεις πληρωμών. Και φέτος είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε παρόμοια παρόμοιου ύψους ε, ποσοστά. Δηλαδή ουσιαστικά το σύνολο των κονδυλίων θα έχει εκτελεστεί από πλευράς προϋπολογισμού. Κατά τη διάρκεια του 2007 είχαμε επίσης ένα υψηλότατο επίπεδο εκτέλεσης. 99,74% σε πιστώσεις ε, πληρωμών και 99,70% σε πιστώσεις ε, πληρωμών. Σε πιστώσεις υποχρεώσεων το πρώτο, πιστώσεις πληρωμών το δεύτερο. Υπάρχει εδώ κάτι και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν επικρίσεις για το ότι δηλαδή δεν γίνονται σωστά οι πληρωμές όσον αφορά τον όγκο των κονδυλίων που μας ζητεί να εκτελεστεί η αρχή του προϋπολογισμού για ένα έτος. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι η απλούστευση, η απλοποίηση. Δράτω με αυτή τη ευκαιρία για να σας εξηγήσω τι είναι αυτό που κάνουμε εμείς στην Γενική Διεύθυνση, σε εμά από πλευράς μας, όσον αφορά την απλούστευση, την απλοποίηση και θα σας αναφέρω γιατί αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόκληση για όλους μας. Όμως η απλοποίηση δεν είναι κάτι που είναι ουδέτερο ή αμερόληπτο όπως μπορεί κανείς ε, να θεωρήσει με μια πρώτη ματιά. Τις πιο πολλές φορές η περιπλοκότητα δεν είναι ένας ε, αυτός σκοπός, αλλά το αποτέλεσμα των διαφορετικών δεσμεύσεων και των, που απορρέουν από τις διαφορετικές ε, διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις και των διαφορετικών ευαισθησιών ε, από πλευράς ε, της πολιτικής αρχής, της αρχής αρμόδιας επί του προϋπολογισμού, των κανόνων που έχουμε θεσπίσει και των αναγκαιοτήτων και αναγκών των όσων συμμετέχουν. Και όλοι αυτοί οι συντελεστές οδηγούν στο να είναι δύσκολο το έργο της απλοποίησης. Μεταξύ των πολιτικών στόχων δίνουμε, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και σε μια παρέκκληση κατά το μέγιστο 2% που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί παρότι έχουμε μειώσει σημαντικά όπως γνωρίζετε το σφάλμα, το ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τα θέματα έρευνας. Από την άλλη πλευρά οι περισσότεροι συμφωνούν στο ότι η έρευνα όπως οποιοδήποτε άλλο κοινοτικό πρόγραμμα πρέπει να απαιτεί μια διαχείριση δημοσιονομική υγιή ώστε οι στόχοι να μπορούν να εκτελεστούν, να επιτευχθούν όμως εκείνο που δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν πρέπει να γίνεται είναι αυτό να είναι ο μόνος στόχος της πολιτικής για την έρευνα. Η πολιτική μας για την έρευνα επίσης έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης επιστημονικής πολιτικής πανευρωπαϊκά στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, αυτή όχι η αντίφαση αφέ αυτής, αλλά μέσα σε αυτή την ισορροπία και μεταξύ των διαφορετικών, να το πω έτσι, ευαισθησιών που υπάρχουν, έχουμε ένα διτό χαρακτήρα. Δηλαδή, σε σχέση με τον ε, εντεταλμένο ε, που πρέπει να αξιολογήσει τα όσα γίνονται από τις υπηρεσίες του για να μπορούν όλες οι ευαισθησίες να ικανοποιούνται. Ενώ πολλές φορές αυτό που βλέπουμε αυτό να συμβαίνει είναι να μην ικανοποιούνται τα πάντα όταν έχουμε διαφορετικές ισορροπίες και ανάγκες. Δηλαδή δεν ε, προσεγγίζει κανείς ε, τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο και έτσι τα πράγματα φαίνεται να μην βρίσκονται στη σωστή ισορροπία όπως θα έπρεπε. Όμως προσπαθώντας να είμαστε το δυνατόν πιο αυτοκριτικοί σε σχέση με τις δράσεις μας θα ήθελα να πω ότι το, πρόγραμμα, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο επέτρεψε να αναπτυχθούν πολλά μέτρα για την απλοποίηση. Ένα μέρος αυτών συνδέονται με το αίτημα του νομοθέτη, δηλαδή ημών, της Ευρωβουλής και του Συμβουλίου και για το θέμα της νομικής βάσης όσον αφορά το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Και το άλλο τμήμα συνδέεται με τις αρμοδιότητες τις δικές μας όταν έρχεται η ώρα της δρομολόγησης όλων αυτών. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία που έχουμε εδώ. Πρώτον, είναι το θέμα του Ταμείου Εγγύησης που μας επέτρεψε να μειώσουμε σε τεράστιο βαθμό τον ε, αριθμό των ελέγχων ex ante. <clears throat> Απαιτούνται πολύ λιγότερα πιστοποιητικά λοιπόν σε σχέση με όσα απαιτούνται στο, στο προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι λοιπόν δυνατό να επιτευχθεί ένα πολύ υψηλό ποσοστό, υψηλότατο ποσοστό εποφελουμένων, πάνω από 80% πιθανότατα, που δεν θα πρέπει ποτέ να δίνουν ή να συντάσσουν κάποιο πιστοποιητικό, διότι το Ταμείο Εγγύησης καλύπτει όλους τους κινδύνους. Τώρα, ο αριθμός των πιστοποιητικών και εντύπων έχει ελαχιστοποιηθεί σε σχέση με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, στο έβδομο που εξετάζουμε. Ο αριθμός ελέγχων εξάντε όσον αφορά τις ικανότητες τις δημοσιονομικές και αυτός ο αριθμός ε, σημαντικά μειώθηκε. Μόνο εκείνη και είναι το ίδιο το κοινοβούλιο όταν το είπε, που το είπε αυτό όταν είχαμε την προηγούμενη συζήτηση. Όταν ζητείτε ένα ποσό πάνω από 500.000 ευρώ, μόνο εκείνοι θα έχουν ένα σύστημα ε, ελέγχου που θα τους διέπει εξάντε. Και αυτό είναι λογικό φαίνεται, διότι κάποιος που υποφελείται από τέτοιο ποσό 500.000 ευρώ είναι ένα σημαντικό ποσό και πρέπει να εξετάζουμε το τι γίνεται. Έχουμε και ένα ενιαίο μητρό συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας ε, για αυτά τα προγράμματα ε, αυτό το μητρό και για όλες τις γενικές διευθύνσεις. Όλοι καταχωρούνται εκεί όσοι συμμετέχουν και έτσι δεν χρειάζεται να συντάσσουν και να υποβάλουν περισσότερα έγγραφα για κάθε συμμετοχή ξεχωριστά. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα το οποίο κάναμε και το οποίο μας κόστισε πολύ ήταν και δαπανηρό ήταν η πιστοποίηση της μεθοδολογίας. Ιδιαίτερα για τις δαπάνες προσωπικού και για τις έμεσες δαπάνες. Με όλα αυτά θα έλεγα ότι θεωρώ ότι θα εισαγάγουμε επίσης ένα στοιχείο απλοποίησης που είναι σημαντικότατο μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Κάτι που κάναμε επίσης είναι ότι απλουστεύσαμε τη διαδικασία για να αλλάξουν οι συμβάσεις ή τα συμβόλαια ή για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Έτσι δύο πράγματα θέλουμε να επιτύχουμε. Να μειωθεί το βάρος το γραφειοκρατικό των εποφελουμένων, αλλά να μειώσουμε και εμείς το γραφειοκρατικό βάρος για μας. Γιατί γνωρίζετε ότι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να υλοποιηθεί με το ίδιο αριθμό στελεχών όπως το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο έχει πολλές ε, δαπάνες ε, για την ε, διαχείριση και μεγάλο όγκο διαχείρισης. Επίσης η περίοδος της διαχείρισης θα είναι μεγαλύτερη ώστε οι επιστήμονες και όσοι εποφελούνται να μπορούν να μην υποβάλουν τόσο συχνά τις πληροφορίες, αυτά τα στοιχεία αυτά προς πληροφόρηση στις υπηρεσίες μας. Μειώσαμε επίσης και τις περιόδους παρακολούθησης. Μειώσαμε όλα αυτά με τρόπο που ο αναγκαίος χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση ενός προγράμματος είναι κατά μέσον όρο 320 ημέρες κατά μέσον όρο που είναι 40 ημέρες ε, μικρότερος αυτός ο χρόνος, αυτό το χρονικό διάστημα από εκείνο που απαιτείται στο έκτο πρόγραμμα ε, πλαίσιο. Αν ακούσετε κάποτε ότι κάποιο σα λέει ότι κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν πιο χρονοβόρο σε σχέση με το 7ο όσον αφορά το 6ο, μια και έχουμε χιλιάδε προγράμματα, μπορεί σε μια περίπτωση να ήταν μεγαλύτερη διάρκεια. Όμω κατά μέσο όρο έχουμε 40 ημέρε μικρότερη περίοδο. Ακόμα και έτσι είναι μεγάλη η διάσταση αυτή η χρονική και θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον χρόνο ακόμα περισσότερο. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε όλες τις αναγκαίες εσωτερικές δράσεις για να επιτύχουμε ώστε όλες αυτές οι περίοδοι, όλη αυτή η χρόνοι να είναι το δυνατόν η βραχύτεροι, η πιο σύντομοι. Κάτι άλλο το οποίο κάναμε είναι η δημόσια διαβούλευση για την απλοποίηση. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε προβλέψει να υποβάλουμε μία πρόταση για την απλοποίηση κατά το πρώτο εξάμεινο του 2010 του επομένου έτους και δεν θέλουμε μόνο τη γνώμη μας να έχουμε και να διατυπώσουμε, θέλουμε να έχουμε και τις απόψεις των διαφόρων εμπλεκομένων που συμμετέχουν και γι' αυτό αυτό που κάναμε είναι δεσμευθήκαμε <clears throat> να κάνουμε μια μεγάλη διαβούλευση με τους όσους συμμετέχουν στα θέματα έρευνας για αυτό το θέμα προωθήσαμε με, με μεγάλο τρόπο, με έντονα αυτή την διαβούλευση, ώστε 3.000 ε, περίπου άτομα έχουν ε, ήδη, ε, έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με αυτά. 30 Σεπτεμβρίου όσον αφορά την ημερομηνία. Όμως δυστυχώς δεν είναι όπως το Ιρλανδικό δημοψήφισμα που μπορεί αμέσως την επόμενη μέρα να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω και να σας αξιολογήσω ποια είναι η γενική άποψη που υπάρχει όσον αφορά την απλοποίηση. <clears throat> Όταν θα, είναι, θα έχει αποκρισταλωθεί αυτή η άποψη για την απλούστευση, για την απλοποίηση, θα γνωστοποιηθεί αμέσως στο Κοινοβούλιο. Τώρα, συγκεκριμένες εξειδικευμένες αξιολογήσεις νομίζω δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά όμως η εντύπωση που έχω αποκομίσει είναι ότι θα μας πούν περίπου το ίδιο και ελπίζω να πούν αυτό ότι υπάρχει σημαντική απλοποίηση και πρέπει να συνεχιστεί η πορεία για την απλοποίηση και στο μέλλον. Αυτό είναι νομίζω το κυριότερο σχετικά. Τώρα τα κράτη, τα κράτη-μέλη όλα συμμετείχαν και είχαν ιδιαίτερα έντονα εμπλακεί στην διαβούλευση η Γερμανία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι κατοχώρες, η Ισπανία <clears throat> καθώς και οι άλλες ε, χώρες σχετικά που συμμετείχαν. Όπως σας έλεγα, έχουμε δεσμευτεί, έχουμε αναλάβει την δέσμευση να προετοιμάσουμε μια ανακοίνωση για την απλοποίηση, για τα θέματα απλοποίησης, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν το δυνατόν ταχύτερα το επόμενο έτος. Και όταν το λέω αυτό, αναφέρομαι κατά τα μέσα, στα μέσα του επομένου έτους ως προς αυτό. Αυτή η ανακοίνωση συμπίπτει και με δύο άλλες σημαντικές, πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που θα κάνει η Επιτροπή. Η μία είναι η τριετής αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και η άλλη είναι η ανακοίνωση για τον ανεκτό κίνδυνο, αποδεκτό κίνδυνο σφάλματος που υπάρχει και που ενέχεται εδώ. Και θα γνωρίζετε ότι για αυτή την ανακοίνωση, για την απλοποίηση, εγώ προσωπικά δεσμεύτηκα και κατέβαλα μεγάλες προσωπικές προσπάθειες. Δεσμεύτηκα ιδιαίτερα ώστε τώρα, σε αυτή τη στιγμή, όταν θα έχουμε τρία χρόνια προγραμμάτων πλαισίου, να βελτιωθούν με τις προσπάθειές μας ακόμα περισσότερο ακόμα περισσότερο αυτά που μπορούν να εξυπηρετήσουν για μια διαχείριση πιο δυναμική, πιο εύκολη, πιο απλή, επίσης και πιο ασφαλή όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ανέφικτα, δεν είναι αδύνατα. Πιστεύω ότι μία από τις τεράστιες δυσκολίες που έχουμε στο πρόγραμμα πλαίσιο είναι το ότι έχουμε υπερβολικά πράγματα που πρέπει να υπαλληθεύονται και υπερβολικά πράγματα που πρέπει να ελέγχονται. Όταν θα έχουμε λιγότερα που πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται, πιο εύκολο θα είναι να υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια απλοποίησης. Πρέπει να είναι σαφές αυτό τα λίγα αυτά πράγματα ή τα λιγότερα πράγματα που θα απομένουν να ελεγχθούν θα πρέπει να ελέγχονται σε βάθος και προσεκτικά και πολύ καλά ώστε οι φορολογούμενοι, οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν ότι τα χρήματα τους, τα χρήματα των φορολογουμένων την χάνουν της καλύτερης χρήσης ε, για ένα σκοπό και στόχο που είναι ιδιαίτερα ευγενής και φιλόδοξος όπως είναι η πολιτική για την έρευνα. Ελπίζω να έχω την τιμή και ενώπιον της Επιτροπής σας ε, στους επόμενους μήνες να προσέλθω και να υποβάλω και παρουσιάσω αυτή την πρόταση, πρόταση για την απλοποίηση ή να συνεισφέρω και να συνεχίσω να επεξηγώ, διότι φυσικό είναι και λογικό ότι από πλευρά τη Επιτροπή θα πρέπει να γίνει αυτή η παρέμβαση. Το τελευταίο στοιχείο επί του οποίου θα ήθελα να κάνω λόγο είναι οι τεχνολογικές κοινέ πρωτοβουλίες, JTI. Όπως γνωρίζετε είναι από τα νέα στοιχεία που έχουμε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Έχουμε πέντε τέτοιες JTI, Artemis, τα καύσιμα των ε, υδρογοναθράκων και διάφορα άλλα σχετικά. Ελπίζω ότι θα ε, υπάρχει αυτονομία αυτών κατά τις επόμενες εβδομάδες, πράγμα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό ώστε να μπορούν να έχουν αυτή την ικανότητα λειτουργικότητας, λειτουργίας ε, για την διαχείριση του προϋπολογισμού τους. Όπως γνωρίζετε, ο Διευθυντής κάθε μιας από αυτές τις κοινέ πρωτοβουλίες τεχνολογιών, JTIs, θα πρέπει να λογοδοτήσει στην Ευρωβουλή για την διαχείριση του προϋπολογισμού των κονδυλίων που είχαν επιμεριστεί και όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα είναι παρούσα και εκπροσωπείται στα governing boards, στα διοικητικά συμβούλια αυτών. <clears throat> Εργαστήκαμε με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν δεν ήταν αυτόνομες, είχαμε διευθυντές ε, και έχοντας ε, ταυτοποιήσει και έχοντας εντοπίσει πλέον διευθυντές ε, από τη στιγμή εκείνη εργαστήκαμε σε ομάδα, ομαδικά μαζί τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είχε ακόμα πλήρως δρομολογηθεί ο αυτόνομος χαρακτήρας του. Συνεργαστήκαμε όμως με αυτόν τον τρόπο μέσα σε ένα ε, ανεξάρτητο πλαίσιο και έτσι ήταν αρκετά παραγωγική αυτή η διαδικασία και οι διευθυντές για την επίλυση του μεγαλύτερου αριθμού των προβλημάτων και θεμάτων που είχαν ε, ανακύψει. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε από την άλλη πλευρά, αυτό που κάνουμε είναι, <clears throat> κάνουμε, επιτελούμε ένα σημαντικό έργο όσον αφορά τις ιδιωτικές δημόσιες εταιρικέ σχέσεις, ΣΔΙΤ, συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΣΔΙΤ, καθώς ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκείνο το οποίο είναι, δεν είναι απόλυτη η ένταξη, όμως έχουμε μία συνεδρίαση ξεκινώντας με τον Επίτροπο Ποτότσνικ και τους ε, επικεφαλείς αυτών των ομάδων και δημιουργήσαμε μια ομάδα ΣΕΡΠΑ, θα έλεγα ομάδα επαφής, ε, ανείχνευσης ε, όσον αφορά το δεύτερο επίπεδο για να λάβουμε υπόψη και να καλύψουμε την, με βάση την εμπειρία που είχε συλλεγεί τις ανάγκες και να δούμε πώς θα έπρεπε να λειτουργούν στο μέλλον και τι θα έπρεπε να γίνει. Ένα σημαντικό θέμα είναι η συμμετοχή των ΜΜΕ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις ΣΔΙΤ, στις συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το άνοιγμά τους προς τον, προς τον έξω κόσμο. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η προσέγγιση ότι αυτές είναι ένας κόσμος αρκετά κλειστός, υπερβολικά κλειστός και στεγανός. Και καταδεικνύοντας το αντίθετο, θα ήθελα να πω το τι έγινε σε σχέση με το Clean Sky. Clean Sky έχουμε 75% των κονδυλίων που άμεσα ε, την χάνουν προς όφελος των ε, εμπλεκομένων και 25% όχι. Γι' αυτό το 25% ήδη ξεκίνησαν 200 προσφορές, 200 προτάσεις. Και έτσι για την χρηματοδότηση περίπου 130 τέτοιων ε, μονάδων έρευνας θα γίνουν σε σχέση με τις συμβάσεις Clean Sky. Αυτό σημαίνει ότι η καταχώρηση σε σχέση, ε, η καταγραφή σε σχέση με τις ε, πιο, ας ε, ολοκληρωμένου χαρακτήρα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η μικρή ίσως πληροφορία που σας προσέφερα είναι χρήσιμη και σας δίνει μια γενική πρόπτικη για το, το πώς έχει εκτέλεση του προϋπολογισμού. Θα είμαστε σε επαφή μαζί σας για οποιαδήποτε πληροφορία θα έχετε ανάγκη να σας παρασχεθεί. Και είμαστε βέβαιοι επιπλέον ότι η πάντα εξαιρετική συνεργασία που διατηρούσαμε μέχρι σήμερα εμείς με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή σας Ήτρε θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια αυτή τη κοινοβουλευτική θητείας και κατά τη διάρκεια τη ανάληψης των πολιτικών πρωτοβουλειών που σχεδιάζουμε για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει ε, σε σχέση με την ε, πανευρωπαϊκή έρευνα. Όπω γνωρίζετε η νέα συνθήκη τη Λισαβόνα μα δίνει μεγαλύτερε ευθύνε και αρμοδιότητε όσον αφορά την έρευνα και ελπίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μα Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Γενική Διευθυντά, για τη διεξοδική αυτή παρουσίαση. Έχουν στήσει αρκετοί συνάδελφοι το λόγο και τους παρακαλώ να λάβουν υπόψη το χρόνο, διότι έχουμε και άλλον έναν προσκεκλημένο στο πρόγραμμα. Σύντομα λοιπόν, όποιος λαμβάνει το λόγο παρακαλώ να επικεντρώνεται σε μία ερώτηση, το πολύ ένα-δύο λεπτά. Πράγμα το οποίο θα μας βοηθήσει βέβαια να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα μας. Ο συνάδελφο κύριος Ρούμπιχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Στο πρόγραμμα βλέπουμε ότι έχετε πολύ καλά ε, σχέδια, την απλούστευση των ε, συμβάσεων, ε, την, τα Μητρώα, Πολύ καλή στόχη λοιπόν, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποιους άλλους περαιτέρω στόχους, περαιτέρω απλούστευση για τις συμβάσεις ή στη διάρκεια της εκτέλεσης. Ξέρω βέβαια ότι έχετε μειώσει στις 320 ημέρες, αλλά υπάρχει στόχος Φερρυπίν για 100 ημέρες ή κάτι άλλο έτσι ουσιαστικό σε προτάσεις. Για δε την χρηματοπιστωτική κρίση θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι σε θέση, αν έχει τη διάθεση να εφαρμόσει στα δικά της, στα του οίκου της την ε, οδηγία την σχετική με τις ε, ληξιπρόθεσμες πληρωμές Late Payment ε, Directive. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της έρευνας και της τεχνολογίας πλήττονται σημαντικά από αυτές τις καθυστερήσεις, τις καταβολές των ε, ποσών. Επίσης στο Caesar, στο EME, ε, e, στο Artemis, στο ENIAC, όπου έχουμε μηδανικές τιμές και στις πληρωμές και στις δεσμεύσεις υποχρεώσεων. Γιατί, γιατί βλέπω αυτό το μηδέν εδώ. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Γιατί δεν υπάρχουν ούτε δεσμεύσεις υποχρεώσεων, ούτε δεσμεύσεις ε, πληρωμών. Και επίσης Στα EITs βλέπω ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, εστιασμός για το Ευρωπαϊκό Τεχνολογίας λοιπόν. Τι καινούριο έχετε να μας πείτε. Ο κύριος πολύ καλό Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βλέπω εδώ ότι ε, ότι υπάρχουν, επισημαίνονται προβλήματα ως προς την ε, περιπλοκότητα των διαδικασιών, ως προς τις βραδιπορίες, την εκτέλεση των προγραμμάτων. Αυτό το θεωρώ ήδη ένα καλό δείγμα ότι σημειώνονται όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα να σημειώσω επίσης ότι υπάρχουν ομάδες επιστημόνων από τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν έχουν μεγάλο ιστορικό θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι νέα κράτη δεν έχουν πολύ μεγάλο ιστορικό παρελθόν. Και φαίνεται ότι αυτά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη και ως προς την αξιοποίηση του επιστημονικού τους, επιστημονικού τους δυναμικού, πράγμα το οποίο θεωρώ λυπηρό και έλλειμμα για ολόκληρη την Ευρώπη. Έχετε κάποιες προθέσεις να βοηθήσετε ώστε στα κράτη αυτά στα οποία δεν υπάρχει πολύ μεγάλη εκπροσώπηση, αν θέλετε, ή εμπλοκή στα επιστημονικά αυτά θέματα, να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης θα πρέπει ασφαλώς να προετοιμαστεί το προσεχές ε, πρόγραμμα πλαίσιο σιγά σιγά. Εγώ για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο κατά την περίοδο της επεξεργασίας του έλαβα υπόψη ε, μελέτες, ε, παρακολούθησα την κατάσταση από κοντά ε, και πρέπει να πω ότι δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος για την διατύπωση του προγράμματος. Από τις μελέτες λοιπόν που θα σας υποβληθούν σκοπεύετε να τις λάβετε υπόψη ή απλώς γίνονται έτσι. Ευχαριστώ Καβάλιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Διευθύντα. Η ερώτησή μου συσχετίζεται με την ε, εκτέλεση σε σχέση με τις χώρες που είναι ένα σημαντικό μέσο για την εμπλοκή της βιομηχανίας στο ΣΔΙΤ. Με τα ίδια τα λόγια του Γενικού Διευθυντή, πολλές φορές είναι ο πιο κλειστός κόσμος σε σχέση με την ε, ε, χρήση των δυνατοτήτων αυτών εδώ σε σχέση με ένα παράδειγμα για την μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να αποκτήσουν ανοιχτό χαρακτήρα. Αυτή η προσπάθεια όμως δεν ήταν η ίδια σε όλες τις ΣΔΙΤ, στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Και είναι δύσκολο αυτό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, πανεπιστήμια, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, μικρές και μεσαίες χώρες, ε, υπάρχουν δυσκολίες. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να εμπλακεί η βιομηχανία και τα κέντρα έρευνας και τα πανεπιστήμια. Και στο σωστό συνδυασμό και με τη σωστή συνεργασία αυτού του τριγώνου της γνώσης που οικοδομούμε θα δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος καινοτομίας και θα χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτό το μέσο που είναι σημαντικό. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν ποια είναι τα σχέδια και τα προγράμματα και τι πρέπει να γίνει ακόμα για να μπορέσει να διασφαλιστεί η ισότητα των ευκαιριών και της πρόσβασης ε, στη διαχείριση των ε, κονδυλίων και στη συμμετοχή και να υπάρξει και χρηματοδότηση και από πλευρά ε, της ε, ιδιωτικής ε, πλευράς και των επιχειρήσεων. Είναι όμως αναγκαίο να έχουμε όλο και περισσότερα τέτοια προγράμματα που θα έχουν ανοιχτό χαρακτήρα και να είναι ανοιχτά για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οντοτήτων των κρατών μελών, διασφαλίζοντας την ισότητα ευκαιριών. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Παστσού παρακαλώ. E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική Διευθυντά, εκτιμώ την επιθυμία σας να πλουστεύσετε τη διαδικασία παροχής οικονομικής βοήθειας για την έρευνα. Ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Να πλουστεύσουμε και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία, των αποτελεσμάτων δηλαδή της έρευνας διότι μόνο αν εφαρμόσετε τα αποτελέσματα της έρευνας στην πράξη, μόνο τότε αυτό γίνεται διαθέσιμο για το κοινό. Γνωρίζω περιπτώσεις όπου μερικές φορές σημαντικές καινοτομίε ή ανακαλύψεις περιμένουν πάνω από ένα χρόνο για να πάρουν προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Και το κοινό περιμένει τα αποτελέσματα πάρα πολύ και δεν χρησιμοποιούνται λεφτά, πράγματα που μπορούν να κάνουν καλό στον κόσμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ μερικές ερωτήσεις. Αν δεν έχετε την απάντηση τώρα, το λέμε αργότερα. Πρώτη, μιλήστε για απλούστευση. Όταν δούμε τα χρήματα που δίνονται στην διαχείριση των προγραμμάτων σε αντίθεση με τα χρήματα που δαπανώνται, θα ήθελα μια αναλογία. Δηλαδή, ας πούμε ξοδεύουμε 100 ευρώ για έρευνα, πόσα ευρώ δίνει η Ένωση για διοικητικά και πόσα ευρώ παίρνουν, πρέπει να ξοδέψουν οι, οι λήπτες των χρημάτων για να τα δαπανίσουν. Θα ήθελα αυτό το πράγμα για να μπορέσω να αξιολογήσω κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η αναλογία, αλλά θα μου ήταν χρήσιμο. Δεύτερη ερώτηση. Είστε ικανοποιημένο με την εστίαση των προσπαθειών για την έρευνα. Ξέρετε, για να πετύχουμε αποτελέσματα πρέπει να πετύχουμε κρίσιμη μάζα. Αν αρχίσουμε να σκορπίζουμε τα χρήματα πολύ, δεν θα πετύχουμε την κρίσιμη μάζα. Θα ήθελα την άποψή σας. Τρίτη ερώτηση. Σε τι βαθμό τα προγράμματα που ξεκίνησαν ως κομμάτι των προγραμμάτων πλαισίου συνεισφέρουν στο εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, πώς αποφεύγετε την επικάλυψη. Ξέρετε ότι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, την, ε, την κοινή έρευνα για τον Αλτσχάιμερ. Πολύ καλή πρωτοβολία. Θα ήθελα να ξέρω, είναι αυτό του ομαλού συστήματος διαχείρισης του προγράμματος πλαισίου ή όχι, πρόεδρος η συνάδελφος Τόμψον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, είχαμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα πριν τα προγράμματα αυτά λειτουργούσαν για τέσσερα χρόνια. Τώρα έχουμε νέα μέθοδο. Πρέπει να ακολουθούν τον προπολογισμό χρονικά. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα. Υπέρ πολλοί ερευνητέ μα εξήγησαν ότι τα προγράμματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνο για τέσσερα χρόνια, θα προτιμούσαν 7 χρόνια. Και όλοι συμφωνήσαμε. Στο μεταξύ όμως, με αυτό το μακρόπνο σχεδιασμό δεν λαμβάνουμε υπόψη την ιστορία, δηλαδή νέα ιστορικά δεδομένα. Γιατί τι γίνεται μετά την οριστικοποίηση, αυτό που συνέβη μάλλον μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος Πλασίου, αυτό έγινε το 2006 και το 2005. Το 2006 όμως ξεκίνησε η κρίση της ενέργειας και του κλίματος. Αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στο νέο πρόγραμμα. Πρόσφατα η Σουηδική Προεδρία ήρθε στην Επιτροπή μας και μας παρουσίασε ένα νέο όραμα, το οποίο θα το δουλέψουν να κοινού την Ισπανική Προεδρία για μια πιο πράσινη Ευρώπη, μια οικολογική οικονομία. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και ρωτώ, πώς μπορεί να έχετε καλά προγράμματα που να λειτουργούν για 7 χρόνια αλλά να είναι ταυτόχρονα και πιο ευέλικτα. Και πώς το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο να γίνει πιο πράσινο σύμφωνα με τις πολιτικές που όπου εμείς αποφασίσαμε με τα νέα πακέτα για την ενέργεια και το κλίμα για τα επόμενα δέκα χρόνια. Πώς τα προγράμματα πλαίσιο θα υποστηρίξουν τη στρατηγική αυτή για την ενέργεια και το κλίμα, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας του 2020. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέρα Ματουρέλ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα, κύριε Σίλβα. Καλώς ήρθατε σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή, σε αυτή την πρώτη σας παρουσία, σε αυτή την κοινοβουλευτική μας θητεία. Θέλω να ευχαριστήσω για τις ε, επεξηγήσεις στην εισήγησή σας που ήταν σαφή και πραγματιστική, ρεαλιστική. Και θέλω να πω ότι Πολλές από τις ερωτήσεις που ε, είχα σκοπό να διατυπώσω με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καλυφθούν. Θα επικεντρωθώ όμως σε δύο ε, θέματα ουσιαστικά. Πρώτα απ' όλα τα JTIs, τις κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες Είχαμε στην έκθεση τα στοιχεία για τα κέντρα έρευνας, πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις και κυρίως μετά από την ανάλυση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των κονδυλίων που όπως είπατε καταδεικνύει ανάγλυφα το τι συμβαίνει. Πιστεύω ειλικρινά και εδώ θα διαφωνούσα μαζί σας ότι ε, και έχουμε ένα πρόβλημα με τις JTIs για το ότι δεν λειτουργούν, για το ότι δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός όπως θα έπρεπε. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε. Γνωρίζετε ότι η ομάδα μου έχει τοποθετηθεί για τους στόχους ε, που έχουν ε, θεσπιστεί. Και με διάφορες ευκαιρίες είπαμε ότι θεωρούμε τα JTIs ως ένα καλό μέσο για να βελτιωθεί η δυνατότητά μας περαιτέρω. Σαφώς ε, βέβαια ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν με τους στόχους ε, που θεσπίστηκαν, αλλά ευθύ εξ αρχής εκφράσαμε και θέσαμε σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή σοβαρές αμφιβολίες για το πώς ε, εξετελούνται τα πράγματα και δρομολογούνται όσον αφορά την χρηματοδότηση, τη συμμετοχή, την διαφάνεια, τον ανοιχτό χαρακτήρα τους και έχετε συνειδητοποιήσει αυτά και κάνετε κάτι για να διασφαλιστεί η επίλυσή τους και δυστυχώς σε σχέση με τα τέσσερα πρώτα επί των οποίων τοποθετηθήκατε, θεωρώ παρόλα αυτά ότι επιβεβαιώνονται δυστυχώς οι ανησυχίες μας και γι' αυτό η ερώτησή μου σε σχέση με αυτό το θέμα. Και ίσως αν θέλετε για να αναφερθείτε να εξηγήσετε περισσότερο και να εξηγήσετε σε σχέση με την πείρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα JTI σας, συνεχίζετε να θεωρείτε ότι αυτή είναι μια βιώσιμη μορφή ε, δράσης θα υπάρξουν περισσότερα JTIs ή στο μέλλον εξετάζετε διαφορετικές ε, μορφές ε, συμμετοχής ε, για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου. Και μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με την αξιολόγηση τους οικονομικούς ελέγχους, τους ελέγχους για τις προσφορές, τις προκηρύξεις και υποβολή προτάσεων και τη συμμετοχή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και για τις, ε, τους γενικούς στόχους. Θέλω να σας πω ότι μου ε, προκάλεσε την προσοχή κάτι το οποίο είδα στην ενδιάμεση αναθεώρηση και που ότι σε σχέση με τους ερευνητές και την έρευνα θα πρέπει να περάσουμε από την πολιτική ελέγχων στην πολιτική εμπιστοσύνης, ενός κλίματος εμπιστοσύνης ερώτηση, τι κάνετε, γίνεται κάτι για τον πολιτισμό και το, την κουλτούρα των, ε, της ε, εμπιστοσύνης. Νομίζω και υπό το πρίσμα αυτό αυτό θα ήταν θετικό και να σας ρωτήσω ή να ζητήσω να σχολιάσετε κάτι για κάποια θέματα. Για παράδειγμα, πώς αξιολογείτε ότι μόνο 10% των ερευνητών που συμμετείχαν σε επιλεγμένα προγράμματα προέρχονται από τα νέα κράτη-μέλη. Να σας ευχαριστήσω για το μέλημά σας ε, για την αύξηση της συμμετοχής γυναικών στα προγράμματα πλαίσιο. Είναι σημαντικό αυτό και καλό. Θα θέλαμε να γίνει μια αξιολόγηση να αποτιμήσετε το ε, Financial Facility και να σας ρωτήσω κάτι επίσης για τις ε, κοινέ προκηρύξεις ε, για το, δυνατότητα αυτής της εταιρικής σχέσης στην έρευνα. Και ολοκληρώνω με αυτό, Πρόεδρε, Ολοκληρώνω και θα ήθελα να πω απλά στον κύριο Σύρβα, ότι τα μέλη της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, και που στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία εμείς που συμμετείχαμε δραστήρια και για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα τον σύνθετο χαρακτήρα, περίπλοκο χαρακτήρα και την δυσκολία όσον αφορά διάφορους, διάφορα θέματα για την εκτέλεση του προγράμματος πλαισίου. Γι' αυτό θέλω να σας ε, ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την εκτέλεση, να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία με την Ευρωβουλή και να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαστε εδώ παρόν στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πολλές σας ερωτήσεις. Η κυρία ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστώ και τον κύριο Ροντρίγκε για την παρουσίασή του και να υποβάλω τρεις ερωτήσεις πολύ σύντομα. Καταρχάς, τα σημαντικότερα κονδύλια για την έρευνα τα διαθέτει το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, όπου έχουν καλές επιδόσεις ορισμένα κράτη συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αυτό, ενώ κάποια άλλη ε, μόνο προσφέρουν χρήματα και δεν απορροφούν για την έρευνά τους. Θα ήθελα λοιπόν να ερωτήσω τι είδους μέτρα σκοπεύετε να προτείνετε έτσι ώστε τα κράτη αυτά τα οποία είναι μόνο καθαροί πλήρωτες να έχουν καλύτερη δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεύτερον, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, που θα πρέπει να συμμετάσχουν, θα μπορούν να συμμετάσχουν υπό το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει να καταβάλουν και οι ίδιες τη δική τους συμμετοχή. Ωστόσο, στην τρέχουσα εποχή είναι δύσκολο να εξασφαλίσει κανείς τη σχετική οικονομική κάλυψη από τις τράπεζες και βέβαια οι επιστημονικές ε, επενδύσεις, οι επενδύσεις στον χώρο της επιστήμης χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς επενδύσεις Υπάρχει κάποια δυνατότητα διευκόλυνσης της πρόσβασης στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και την ερώτηση αυτή την ε, υποβάλλω, διότι είναι αναγκαίο πιστεύω να έχουμε περισσότερες ε, επενδύσεις στις καινοτόμους, στον τομέα της καινοτομίας, εκεί ακριβώς που υπάρχει λιγότερη ε, ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρε, είμαι νέο μέλος, νέος ευρωβουλευτής και υπό αυτή την ιδιότητα μια ερώτηση θα ήθελα να διατυπώσω. Θα έλεγα, δεν είναι μόνο το ότι δεν έχω αρκετές πληροφορίες. Έχουμε και κάποια νέα στοιχεία τα οποία γνωστοποιήθηκαν για την αξιολόγηση και, για τα, και τα στοιχεία δείχνουν, λένε ότι 25.000 ε, αιτήματα διατυπώθηκαν, 5.000 εγκρίθηκαν 1170 προσφυγές έγιναν ή παράπονα και εγκρίθηκαν κάποια από αυτά. Και φυσικά οι φορολογούμενοι θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς για ποιο σκοπό δαπανώνται τα κονδύλια των φορολογουμένων. Θέλουν όμως επίσης να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας και ποια επιτυχία συνεισφέρουν αυτά τα προγράμματα. Επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι κάποια κοινωνικά ωφέλη και οικονομικά ωφέλη πρέπει να ε, επιτυγχάνονται. Είναι αυτό σημαντικό και θα ήθελα να ρωτήσω ποια μέσα, ποια εργαλεία έχετε για να αξιολογήσετε Πώς αξιολογείτε αν εκτελέστηκε ικανοποιητικά ένα πρόγραμμα ή αν ε, ε επετεύχθη όπως ε, απαιτεί η σωστή ε, εφαρμογή του. Και αντίστοιχε εκθέσεις θα έπρεπε να συντάσσονται σπανιότερα από ό,τι στο παρελθόν. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι έχετε τα αναγκαία μέσα στη διάθεσή σας και τα εργαλεία να αξιολογήσετε το follow-up, τη συνέχεια, το όφελος που επιτυγχάνετε και συνοδευτικά να δώσετε πληροφορίες σχετικά, διότι οι φορολογούμενοι κατά πρώτο λόγο ενδιαφέρονται να τα μάθουν όλα αυτά. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ο κ. Χατζημαρκάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγηση βάσει των οποίων διατίθενται τα κονδύλια, στα οποία αναφέρθηκε ο και ο Και θα ήθελα να μου πείτε αν αποκλείεται ορισμένη τομή της έρευνας... να ε, θεωρηθεί ότι δεν έχουν απόδοση ή δεν έχουν αναγνωριστημότητα. Την έννοια ότι δεν δικαιολογεί επαρκώς την ε, χορηγία ο ε, υπεύθυνο του προγράμματο, εκείνο που ζητεί τη χρηματοδότηση, δηλαδή, ότι θεωρείται ότι δεν είναι ικανοποιητικό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε πολλέ ερωτήσει και ελπίζω όσο το δυνατόν πιο εστιασμένα να δώσετε και τις απαντήσεις σας, χωρίς αυτό βέβαια να είναι εύκολο καθήκον που σας αναθέτω. με την άνεση σας φυσικά, αλλά ή δυνατόν να απαντήσετε στα πιο σημαντικά. Κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολο να απαντήσω σε σχέση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, την Επιτροπή που γνωρίζει απόλυτα το έργο και θέτει άμεσα ερωτήσεις στον Γενικό Διευθυντή. Είναι απλό. Στην, στο, στο web site της Γενικής μας Διεύθυνσης μπορεί κανείς να απευθυνθεί και να αντλήσει στοιχεία. Θα το κάνω όμως εδώ άμεσα. Δεν είμαι ε, ένα άτομο το οποίο να ε, με ενοχλεί το να είμαι ε, σε σχέση με την δυνατότητα χορήγησης απάντησης σε αυτά τα θέματα στα ισπανικά όλας άμεσα. Η πρώτη για το ερώτημα το οποίο έγινε. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περαιτέρω το θέμα των προθεσμιών, να πληρώνονται σε 30 μέρες, να υπάρχουν πληρωμές είναι αρκετά περίπλοκο το να πληρώνει κανείς σε 30 μέρες. Ακόμα και έτσι όμως το καταφέρνουμε, το πετυχαίνουμε σε ένα πρόγραμμα όπου υπάρχει ταχύτατη δυνατότητα ε, χορήγησης, ε, ε, εκτέλεσης πληρωμών. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με αυτά τα παραδείγματα να προχωρήσουμε και να τα μιμηθούμε σε άλλες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι να επισπεύσουμε τις πληρωμές είναι ένα μόνιμο μέλημα. Διαρκώς βελτιώνουμε τα πράγματα, διαρκώς. Τώρα Τώρα για το ερώτημα αν ε, υπάρχει αυτή η βελτίωση, όχι μόνο να έχουμε το θέμα των πληρωμών σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να είμαστε ικανοί, να είμαστε πάντα αποτελεσματικοί για τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων και πιστώσεις ε, πληρωμών. Ναι, έκανα λόγο και μίλησα γι' αυτό και για την εκτέλεση και των πιστώσεων υποχρεώσεων και τις, τις πληρωμών και για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας ε, δεν συμμετέχει στην ε, γενική μας ε, διεύθυνση. Θα προτιμούσα να θέσετε αυτό το ερώτημα στον συνάδελφό μου που θα προσέλθει και για τα JTIs πολλοί από εσά αναφέρθηκαν σε αυτό και θα προσπαθήσω υστερότερα να απαντήσω αυτό το σημείο. Σαφώς υπάρχει η δέσμευση να βελτιώσουμε και σας δίνω τη δέσμευσή μου για τη βελτίωση αυτή. Από την στιγμή που ανέλαβα αυτό το αξίωμα μειώσαμε τις ε, προθεσμίες, τις διορίες και θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Μου θέσατε εσείς ε, και κάνατε λόγο για τα νέα κράτη-μέλη. Για μένα πάντα ήταν ε, μεγάλο μέλημα, ιδιαίτερα έντονο, ώστε στο πρόγραμμα πλαίσιο να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα πολύ απλό λόγο διότι αν δεν υπάρχει αυτή η εκπροσώπηση θα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρέπει να διατηρούμε το δι, διτό στοιχείο, τον εξαιρετικό ε, χαρακτήρα όσον αφορά τι επιδόσει αυτού του προγράμματο πλαισίου που είναι η πρόσθετη αξία που δημιουργούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να κάνουμε και ό,τι περνάει από το χέρι μα για να έχουμε μια εκπροσώπηση κάθε φορά υψηλότερη. Αλλά μην ξεχνάμε και ένα άλλο θεμελιώδε στοιχείο, ότι υπάρχουν άλλα στοιχεία και εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στα διαθροτικά κονδύλια. Τα διαθροτικά κονδύλια έχουν μεγαλύτερο ποσό για τέτοιες δραστηριότητες έρευνας από ότι το ίδιο το πρόγραμμα πλαίσιο. Έχουμε ε, περισσότερα από 58 ε, εκατομμύρια ε, ευρώ που έχουν καταχωρηθεί σε, στα διαρθρωτικά κονδύλια. Μεταξύ της συνέργειας αυτών των ε, του προγράμματος πλαισίου και των διαρθρωτικών κονδυλίων μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Είμαστε πραγματικά ευθυγραμμισμένοι ώστε να πετύχουμε τη συνέργεια και τις επιπτώσεις από συνεργειακές δράσεις. Η κυρία Καρβάλιο έκανε λόγο για τα JTIs και ίσως ε, στην απάντηση που θα της δώσω θα πω τα θεμελιώδη τα οποία εγώ πιστεύω σε σχέση με τα JTIs. Τα SDIT είναι η πιο, ας το πω έτσι, ε, τολμηρή πλευρά και συνιστόσα όλων των δράσεων στο πρόγραμμα πλαίσιο υπό το δημοσιονομικό χρηματοδοτικό τμήμα το πιο αναγκαίο όσον αφορά τη δημιουργία καινοτομίας και τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης. Πρέπει να συνδυάσουμε και να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και να παίξουμε να διαδραματίσουμε ρόλο με αυτά τα στοιχεία. Και με το, το θέμα του κινδύνου του δημοσιονομικού που είναι μεγαλύτερος όσον αφορά το European Research Council, από την άλλη πλευρά έχουμε την ανάγκη δημιουργίας καινοτομίας. Και αυτή την ανάγκη την αναφέρει στην χορήγηση απαλλαγής ε, που έδωσε η Ευρωβουλή στο τελευταίο έτος. Ζητείτε για κάθε Joint Technology Initiative να υπάρχει ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο κεφάλαιο στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων από πλευρά μα. Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει λοιπόν ότι είναι αναγκαίο αυτό σε μεγάλο βαθμό και γνωρίζουμε ότι εμπλέκονται μεγαλύτεροι κίνδυνοι και είναι επισφαλέστερο αυτό από ότι άλλε δράσει. Πρέπει να συνδυάσουμε αυτό σε σχέση με τα ευαίσθητα αυτά σημεία για τα οποία σας έκανα λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε, να συνεργαστούμε με τους διαφορετικούς εμπλεκομένους με τη μέγιστη διαφάνεια. Ήδη σας είπα ότι έχουμε μία ομάδα με όλα τα JTIs. Εγώ είμαι προεδρεύω ίδιος και ανταλλάσσουμε εμπειρίες σε αυτή την ομάδα για να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε στο μέλλον για τις νέες JTIs και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα καινοτόμο αυτή τη στιγμή αλλά θα υπάρξει κάτι και αν είναι δυνατόν να βελτιωθεί κάτι για τις ε, JTIs, ε, να υπάρξουν χειροπιαστές βελτιώσεις. Ένα θεμελιώδες στοιχείο που πρέπει να έχουν οι JTIs είναι ο ανοιχτός χαρακτήρας και η πρόσβαση για όλους. Και ανέφερα την περίπτωση των Clean Skies με μεγαλύτερη προσπελασιμότητα, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αυτή που είχε αρχικά υπολογιστεί και αυτό πρέπει να προαχθεί σε όλες αυτές τις δράσεις. Οι προκηρύξεις πρέπει να είναι ανοιχτές και διάφανες με τον ίδιο τρόπο όπως Ανοιχτές και διάφανες είναι οι προκηρύξεις για άλλες δράσεις που ε, ε, καλύπτονται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αναφερθήκατε εσείς στο, στα θεμελιώδη στοιχεία. Ποια είναι τα θεμελιώδη στοιχεία εδώ. Είναι τα θεμελιώδη στοιχεία όλου του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, η προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η εφαρμογή, εκτέλεση των αποτελεσμάτων με τον βέλτιστο τρόπο. Έτσι, με συγκρίσιμο τρόπο, συγκρίνοντα μεταξύ των κρατών μελών, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν καθυστερήσει. Αυτέ όμω οι πρωτοβουλίε δεν βρίσκονται με σαφήνεια μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα πλαίσιο. Βρίσκονται περισσότερο μέσα στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα. Του Ευρωπαϊκού Χώρου για την έρευνα που με τη νέα συνθήκη τη Λισαβόνα θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Και δεν έχω πρόβλημα όποτε θέλετε να ξαναέρθω εδώ στην κοινοβουλευτική σας επιτροπή για να ξανακάνω λόγο για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στον Ευρωπαϊκό χώρο για την έρευνα πρωτοβουλίες που από κοινού συμμετέχουν σε αυτές τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ε, Ένα άλλο στοιχείο θεμελιώδες που ανέφερε ο κύριος Λάμπερτς. Πόσα είναι αυτά τα οποία διατίθενται στα, πειραματικά εργαστήρια τι γίνεται με τα κονδύλια. Εγώ από πλευρά μα έχουμε ένα βάρος για τη διαχείριση που έχουμε αναλάβει 6% σε σχέση με τις δαπάνες. Δεν φτάσαμε ποτέ σε αυτό το 6%. Βρισκόμαστε στο 4% και καμιά φορά και λιγότερο. Όμως από την άλλη πλευρά εκείνο που είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω εγώ ίδιος αυτή τη στιγμή είναι τι γίνεται σε σχέση με το γραφειοκρατικό βάρος και την επιβάρυνση που ε, συνοδεύουν κάθε σχέδιο. Πιθανώς έχουμε κάποια μεγάλη επιβάρυνση Είμαι όμως βέβαιος σε σχέση με τις δαπάνες για τα κέντρα έρευνας είναι μεγαλύτερα τα κονδύλια από ότι αυτά τα οποία εμείς δαπανούμε. Και λογικό είναι, αν θα μπορούσε αυτό να επανορθωθεί, να διορθωθεί θα ήταν εξαιρετικό. Πρέπει να έχουμε όμως πολύ απλούστερους κανόνες και σαφέστερους κανόνες, διότι το περισσότερο γραφειοκρατικό στοιχείο, το μεγαλύτερο γραφειοκρατικό στοιχείο είναι ρήτρε και διατάξεις για την εφαρμογή των κοινών κανόνων. Τη στιγμή που αλλάξουμε ένα μέρος αυτών των κανόνων θα είναι πιο απλό. Θα είναι πιο απλό να ελέγξουμε αυτές τις δράσεις αφενός. Και από την άλλη πλευρά θα είναι πιο απλό να έχουμε και την αναχέτηση, την αντιμετώπιση των ε, ε, βαρών που επιβαρύνουν τα κέντρα έρευνας. Ο σωστός στόχος πρέπει να, να καλυφθεί. Να είμαστε με σωστή στοχοθέτηση όταν υποβάλλονται οι προκηρύξεις. Ε, ακούστε γι' αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε ένα στοιχείο πάρα πολύ αξιόλογο. Κάθε χρόνο έχουμε ένα πρόγραμμα εργασίας. Σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας κάνουμε μια μεγάλη κοινή διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση και σε σχέση με τα κράτη-μέλη για το ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι κάθε ενός από τους ε, τομείς αυτούς στην Ευρώπη. Όμως επίσης έχουμε και το ίδιο το πρόγραμμα που ο πρόεδρος ε, Μπαρόσο ε, ξεκίνησε και στο οποίο αναφέρεται ότι έχουμε και κάποια σημαντικά στοιχεία. Πώς πρέπει να διαμορφωθεί το πρόγραμμα για την έρευνα. Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα ακριβώς έχει αυτά τα μέσα για την υλοποίηση αυτών των στόχων και προτεραιοτήτων. Έχουμε λοιπόν σαφή στοχοθέτηση και προτεραιότητες. Με ρωτήσατε και μου είπατε πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να είναι πιο ευδιάκριτη και πιο πράσινη η πολιτική για την έρευνα. Είναι αυτονόητο και λογικό ότι πρέπει να γίνει και θα γίνει πιο πράσινη και θα πρασινίζει κάθε χρόνο. Διότι θα έχουμε μια κοινωνία χαμηλού ποσοστού άνθρακα. Και έτσι για τις προκηρύξεις εγκάρσιου χαρακτήρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έχει στοιχεία τα οποία κάθε χρόνο με αυτόν τον τρόπο ε, εναλλάσσονται για την επίτευξη των στόχων. Τώρα, η συμπληρωματικότητα όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα και τις επικαλύψεις. Για το πρόγραμμα πλαίσιο που έχει συγκεκριμένη αξία πρέπει δύο πράγματα να υπάρχουν. Η πρόσθετη αξία όσον αφορά τι δράσει των κρατών μελών και από την άλλη πλευρά να αποφύγουμε επικαλύψεις. Όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί και πραγματιστές. Υπάρχουν πολλές επικαλύψεις μεταξύ των πολιτικών έρευνας των 27 κρατών μελών σε σχέση με τις επικαλύψεις του 7ου προγράμματος πλαισίου και του τι γίνεται από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα παράδειγμα που πάντα αναφέρεται ότι δηλαδή σε σχέση με το ε, βακτηρίδιο αυτό το οποίο βρίσκεται στα, στα πουλερικά ότι το ίδιο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού αν είναι δυνατόν θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί έχουμε και κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται για να έχουμε ένα κοινό προγραμματισμό μεταξύ των κρατών μελών και σε σχέση με τις δράσεις και πληρωμές. Είναι δύσκολο, κυρίως γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο. Όμως κάθε φορά που κάνει κάποιος κάτι για πρώτη φορά είναι ιδιαίτερα δυσχερές το εγχείρημα. Εσείς ε, αναφέρατε ότι όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχουν τα προγράμματα πλαίσιο τόσο καλύτερο. Πιστεύω ότι αυτό το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο που έχει 7 έτη ε, διάρκεια, σύμφωνα με τι δημοσιονομικέ προοπτικέ, μα επιτρέπει πολύ περισσότερο περιθώριο ελιγμών για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην ε, ίδια την πραγματικότητα. Έχει αλλάξει όμω ο ίδιο ο κόσμο αυτά τα τελευταία 7 ε, χρόνια. Όταν είχα έρθει το 2006 να μιλήσω μαζί σα για το πρόγραμμα πλαίσιο, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, οι προτεραιότητε ήταν διαφορετικέ. Άλλα θέματα απέρευσαν και πρέπει να προσαρμοστούμε ώστε να είμαστε αρκετά ευέλικτοι στο πρόγραμμα αυτό για να μπορούμε να προσαρμοστούμε στην ίδια την πολιτική πραγματικότητα και στην ίδια την οικονομική πραγματικότητα με τις προσαρμογές μας. Η κυρία Ριέρα τα, τα ρωτάει όλα δεν ε, γνωρίζω μήπως θα έπρεπε να προσκαλέσω σε δείπνο για να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που ε, μου έθεσε και να μπορέσω να τα καλύψω όλα. Για το Joint Technology ε, Initiatives πρέπει να συνδυάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά τη συμμετοχή που πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους εμπλεκόμενους των JTI, στην ελαστικότητα των μηχανισμών που πρέπει να διασφαλίζεται, πιθανότατα η νομική μορφή για το community bodies θα πρέπει να είναι το έργο που πρέπει να μας απασχολήσει και κάνουμε πραγματικά προβληματιζόμαστε για το μέλλον, τι πρέπει να γίνει μέσα στο πλαίσιο των ε, κοινών αυτών δράσεων που είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συνδυάσουμε τις, ε, το προϋπολογισμό από πλευράς, ε, τα κονδύλια από πλευράς ε, του ιδιωτικού τομέα και τα δημόσια κονδύλια από πλευράς των φορολογουμένων τις κρατικές δράσεις. Τώρα, διατυπώσατε μια άλλη ερώτηση κυρία Ριέρα, μια στιγμή. Λυπούμε, δεν δεν είναι το 10%, το 10% είναι για τα νέα κράτη-μέλη, για την εκπροσώπηση. Εντάξει, το 10% για τα νέα κράτη-μέλη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμως ότι έχουμε δημιουργήσει και μεγάλες εκδηλώσεις όπως και με την Τσεχική Προεδρία για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε για να υπάρξει συμμετοχή μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι όσο μεγαλύτερη σημασία δίνει ένα κράτος στην πολιτική έρευνας από πλευράς ε, του όσο περισσότερα δαπανά στον εθνικό προϋπολογισμό για την πολιτική έρευνα σε ένα κράτος, τόσο καλύτερα αποτέλεσμα επιτυγχάνονται και όσον αφορά τη συμμετοχή στο κοινοτικό πρόγραμμα για την έρευνα. Διότι είναι πολύ ανταγωνιστικά προγράμματα και πρέπει να είναι ανταγωνιστικά και πρέπει να έχουν αυτό το χαρακτήρα. Γι' αυτό όσο πιο προετοιμασμένη και προπονημένη είναι μια χώρα, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι. Τώρα, για την δυνατότητα για το ε, Risk Management Facility, για την αντιμετώπιση κινδύνων, υπάρχει εδώ τεράστιο δυναμικό καινοτομία. Είναι η πρώτη φορά που σε σχέση με μια τράπεζα υπάρχει η εξέταση αυτού του κινδύνου για την ε, χρηματοδότηση. Και εδώ θέλω να ζητήσω να υπάρξει υποστήριξη. Ξεκινάμε την ιδέα ότι μέσω των, της χρηματοδότησης ε, για την ε, έρευνα δεν έχουμε μόνο τις κρατικές τράπεζες, πρέπει και τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο κόσμος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να κινητοποιηθεί, να τους πούμε ότι είναι καλή πρωτοβουλία αυτή και έχει θετικά ωφέλη και για αυτούς. Τώρα, όσον αφορά κάθε φορά όλο και περισσότερο τις δράσεις που ακολουθούμε για τις κοινέ προκηρύξεις διότι δύσκολο είναι να υπάρξει ε, ανάμιξη δύο διαφορετικών συνιστοσών ε, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Όμως όλο και περισσότερο πρέπει να προχωράμε σε θέματα που θα συνδέουν το περιβάλλον με θέματα ενέργειας, ενεργειακά και με άλλες προτεραιότητες και είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι για το τι πετυχαίνουμε. Η κυρία Τικάου για μέτρα ώστε όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν και να υποφελούνται. Λοιπόν, ακούστε, νομίζω έχει γίνει κάποια παρέμβαση σχετικά ήδη και θεωρώ ότι είναι αθεμελιώδους σημασίας. Επισκέφθηκα τα, κέντρα των κρατών μελών εκτός από ένα και θα το ε, επαναλάβω για άλλη μια φορά. Υπάρχουν θεμελιώδη στοιχεία εδώ. Να δεσμεύσουμε τη συνέργεια των διαθροτικών ταμείων με τις δράσεις του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Έχει θεμελιώδη ρόλο να διαδραματίσει αυτός ο συνδυασμός, ο συγκερασμός αυτών των δύο δυνατοτήτων. Τώρα, σε σχέση με τον συνδυασμό αυτό, συνδέεται με αυτό που είπα. Είναι θεμελιώδες να ευαισθητοποιήσουμε ιδιωτικούς, ε, ε, τον ιδιωτικό τομέα για αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Και εδώ έχουμε και το ε, τομείς όπου για παράδειγμα όσον αφορά και τις ε, οικοδομές μπορεί να είναι ε, θετικός. Ποια είναι η επιτυχία των πρωτοβουλειών αυτών ρωτήσατε. Πώς μπορούμε να τα μετρήσουμε όλα αυτά στις επιπτώσεις τους. Λοιπόν ακούστε υπάρχει ένα τμήμα που προσπαθούμε να μετρήσουμε τώρα στην αξιολόγηση του έκτου και στο μέλλον στην αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Προφανώς είναι δειγματοληπτικές αυτές οι, αξι... αξιολογήσεις. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εξάντε και εξ post γίνονται πάντα. Δεν μπορούμε εξ να γνωρίζουμε εκ προημίου ποια θα είναι τα αποτελέσματα ενός πακέτου μιας δράσης για την έρευνα. Και είναι επίσης και διαφορετικό αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε σε σχέση με, κάποιο, ε, με κάποια τέτοια πρωτοβουλία έναντι μιας άλλης. Όταν ε, έχουμε μια επιχορήγηση και υποστήριξη για μια δράση ε, προφανότατα το επίπεδο κινδύνου είναι λόγω του χαρακτήρα του ίσως ε, μεγαλύτερη. Όταν έχουμε μία δράση clean sky έχουμε ένα κινητήρα καθαρότερο. Γι' αυτό έχουμε αυτή την, ε, αυτόν τον τίτλο. Οι Joint Technology Initiatives πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα απριόρι που θα είναι καθαρότερο το αποτέλεσμα σε σχέση με, το, με τις ε, εκπομπές ρήπων και να είναι θετική η δράση για το περιβάλλον. Εσείς κύριε ρωτήσατε, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά σας και έχουμε έρθει σε επαφή. Χατζημαρκάκης μάλιστα. Λέτε λοιπόν τι πρέπει να γίνεται όταν δεν έχουμε αποτελέσματα. Να σας επαναλάβω αυτό, κάπως, αυτό το οποίο είπα πιο πριν. <clears throat> Πώς θα πρέπει σε σχέση με τα αποτελέσματα από την θετική ε, επιστημονική δράση να ζητάμε να υπάρξει η καλύτερη απόδοση. Και όταν έχουμε τα Joint Technology Initiatives πρέπει να ζητάμε πάντα να υπάρχει output διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι η διαδικασία επιλογής που γίνεται απριόρι έχουμε ήδη επιλέξει εκ προημίου τι είναι εκείνο το οποίο επιθυμούμε να πετύχουμε και έχουμε σαφέστερα αποτελέσματα. Τώρα, ποια είναι εκείνη η ερώτηση την οποία δεν έχω καλύψει και που θα έπρεπε να απαντηθεί. Σε σχέση με την εκπροσώπηση, χαμηλή εκπροσώπηση των νέων κρατών μελών από τα νέα κράτη-μέλη. Όχι, σε αυτό το δείπνο που είπατε ότι θα προσφέρατε για να απαντηθούν τα υπόλοιπα, εκεί θα αναφερθεί. Λοιπόν, για την εκπροσώπηση των ε, νέων κρατών μελών. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο έκανε ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό και είχα ευκαιρία να το, να το αναφέρω σε κάποιους από εσάς. Άλλαξε το ποσοστό τελικά. Το staffing grants, των staffing grants, διότι έχουμε εδώ μεγαλύτερη κατανομή πανευρωπαϊκά θα πρέπει να διατηρήσουμε σε όλα τα ποσά, σε όλα τα κονδύλια του 7ου προγράμματος πλαισίου ένα στοιχείο ε, ε, θα έλεγα εξαιρετικών επιδόσεων ε, και που αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζει αυτές τις δράσεις πανευρωπαϊκά. Διότι αν δεν γίνει αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε φιλόδοξο πρόγραμμα πλαίσιο και έτσι θα πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να μπορούν να εκπροσωπούν με αυτό το χαρακτήρα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Γραμματέα για την απάντηση πολλών διαφορετικών ερωτήσεων. Θα είμαι σύντομος. Σίγουρα προ, ε, προφανώς στο μέλλον θα ξανασυζητήσουμε αναμεταξύ μας, διότι είναι σημαντικό έργο και για μας το θέμα του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, αλλά και για το θέμα του πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.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 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf äh, in unserem Kreise erneut. Ήθελα ανάμεσά μα να ξαναχαιρετήσω για αυτή την κοινοβουλευτική θητεία όμω για πρώτη φορά, ενώ τον είχαμε επανειλημμένα στο παρελθόν, τον Λόρδο Τζον Μόγκ, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια. Στην επόμενη κοινο, στην ε, κοινοβουλευτική θητεία που πέρασε είχαμε πολλές φορές επαφές, ήταν έντονες οι συζητήσεις που είχαμε. Χαίρομαι που μπορώ να σας χαιρετήσω και να σας προσφέρω την ευκαιρία σύντομα να κάνετε την παρέμβασή σας και στη συνέχεια αγαπητοί ευρωβουλευτές εσείς ως μέλη θα έχετε την ευκαιρία να διατυπώσετε ερωτήσεις. Παρακαλώ Λόρδε Τζον Μαγκ. Uh, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, καταρχήν σας ευχαριστώ για την ευκαιρία στην αρχή της νέας περίοδου στο Κοινοβούλιο να σας μιλήσω. Καταρχήν όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πρώην βουλευτές που είναι παρόντες και τα νέα μέλη για την άριστη και το τονίζω άριστη υποστήριξη που είχαμε στις συζητήσεις μας για το τρίτο πακέτο. Είχαμε πάρα πολύ συνεργασία και με τους συζητητές, πάρα πολύ στενή συνεργασία με τους ρυθμιστές έτσι ώστε να δώσουμε ανεξάρτητη συμβουλή στους συναδέλφους σας και εμείς από την πλευρά μας να αναπτύξουμε μερικές πτυχές του πακέτου όπου το Συμβούλιο ήταν κάπως διστακτικό στο να κάνει προτάσεις. Αυτό δείχνει και το άνοιγμα που έχουν δείξει και οι ρυθμιστές. Δηλαδή εξακολουθούμε να σας πληροφορούμε, παραδείγματο χάρη, τονίζοντας την ανάγκη του χαρακτήρα του υπόλογου των ρυθμιστών. Γιατί έχουμε περισσότερες εξουσίες και μεγαλύτερη ανεξαρτησία, αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε κάτι πέραν παντός ελέγχου. Αυτό αφορά και τις κυβερνήσεις, οι οποίες δίνουν εξαρτησία, αλλά απαιτούν έλεγχο. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το Κοινοβούλιο. Ένα άλλο σημείο είναι τα μέτρα για τον καταναλωτή, τα οποία τόνισε ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, το λιανεμπόριο. Εμείς ως παρατηρητές στη διαδικασία της συναπόφασης για την απόφαση Μαρόνι που δεν μπλοκάρισε την πιο φιλόδοξη κίνηση των εισηγητών να δώσουν περισσότερες εξουσίες στη νέα υπηρεσία αυτή. Αυτά αφορούν το παρελθόν. Θα ήθελα όμως να αποδώσω φοροτιμή στο τι έγινε στο παρελθόν. Δεύτερο, τώρα έχουμε μια διαδικασία που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. 18 μήνες μετά την έγκριση του πακέτου πρέπει να γίνει η εφαρμογή. Αυτό είναι ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, η Κομισιόν πρέπει να φροντίσει να συμβεί οι, εθνικοί ρυθμιστές να έχουν περισσότερη ανεξαρτησία. Εμείς ως εθνικοί ρυθμιστές πρέπει να προετοιμαστούμε για τη σύσταση της νέας υπηρεσίας. Πρέπει να βρωθεί η διευθυντής. Έχει γίνει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Τι δουλειά θα κάνει η υπηρεσία, πρέπει να προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Θα αναφερθώ σε αυτό. Εμείς λοιπόν ως ρυθμιστές με την συνεργατική συμφωνία που έχουμε στο Βέλγιο, ΣΥΑΡ και το ΕΡΓΕ που είναι το όργανο που έχει συστηθεί από την Κομισιόν <clears throat> θα προετοιμαστούμε πρώτον να γίνει υπηρεσία. Χρειάζεται έδρα. Θα την αποφασίσει το Συμβούλιο, μάλλον το Δεκέμβριο μεταξύ τριών χωρών. Χρειάζεται διευθυντή. Τρίτον, χρειάζεται μια δομή που θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο από τα κράτη-μέλη και εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Ένα Συμβούλιο Ρυθμιστών, αυτό είναι το νέο στοιχείο της υπηρεσίας, Καταρχήν λοιπόν πρέπει να συσταθεί η υπηρεσία, ελπίζουμε το Μάρτιο, να έχουμε την Επιτροπή των Ρυθμιστών, περίπου τότε και αυτή, για να είμαστε έτοιμοι, φροντίζουμε τώρα να έχουμε τους κανόνες διαδικασίας. Μπορεί να φαίνεται γραφειοκρατική, αλλά σας διαβεβαιώνω θα είναι αποτελεσματική. Πρέπει να αποφασίσουμε στους κανόνες αυτούς πώς θα γίνει η ψηφοφορία, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος αντιπρόεδρος, τι εξουσίες θα έχουν, πώς θα τις ασκούν. Πριν γίνει η υπηρεσία αυτή, με το που θα γίνει η υπηρεσία, όπως σας είπα το Μάρτιο, μάλλον, θα αρχίσει η δουλειά. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, η συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες έχουν μεγαλύτερες εξουσίες, μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Για κάποιες χώρες η διαφορά είναι μικρή, όπως για το Ηνωμένο Βασίλειο. Για άλλες χώρες ο ρυθμιστής ήταν τμήμα του Υπουργείου, στο οποίο δούλευε. Τώρα φεύγει από το Υπουργείο, γίνεται ανεξάρτητος, με εξουσίες αν εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία. Επίσης, δεν πρέπει να έχουμε κατακαιρματισμό των εθνικών προσπαθειών. Η υπηρεσία θα τα συντονίζει αυτά. Ο κινητήρας θα είναι οι κανόνες που θα οριστούν στην νομοθεσία. Και λέω κινητήρας διότι χρειαζόμαστε λεπτομερείς κανόνες έτσι ώστε όλοι όσοι παίρνουν μέρος, οι χώρες, οι επιχειρήσεις που θα λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο αυτό, να ξέρουν τι κάνει ο καθένας σε έκτακτη ανάγκη ή σε συνεργασία. Τους κανόνες αυτούς τι κάνουμε. Έχουμε δύο πιλότους, το ένα στο αέριο, το ένα στον ηλεκτρισμό, με δύο νέα όργανα, με τα TICS, ένσο E και ένσο G είναι τα αρχικά για ηλεκτρισμό και αέριο και συνεργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε σωστή λειτουργία έτσι ώστε θα έχουμε την υπηρεσία να μπορούμε να δούμε κατά πόσο τα πράγματα έχουν οριστεί σωστά. Πολύπλοκα πράγματα αυτά. Τα περισσότερα είναι νομικά. Γι' αυτό η προσπάθεια θα αναπτυχθεί σε αυτή την προκαταρκτική φάση. Τώρα κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο και τα θέματα καταναλωτών κυρίως. Το μεγάλο θέμα της, του ασφαλούς εφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας της ενεργειακής αγοράς σε επίπεδο ατομικό ήλιαν εμπορίο. Το Κοινοβούλιο μας έριξε το γάντι και μας προκάλεσε πολλή δουλειά στους ρυθμιστές. Το φόρουμ του Λονδίνου, όπως το λέμε, ανάλογα με το φόρουμ της Φλωρεντίας και της Μαδρίτης, την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε τέτοια θέματα που σας αφορούν και εσά και εμένα ως ανεξάρτητους επιμέρους καταναλωτές. Πάμε χάρη η τιμολόγηση της λογαριασμού ε, λογαριασμούς ενέργειας. Όταν υπάρχει ένα παράπονο του καταναλωτή, πώς λύνεται. Μια μελέτη της αγοράς που θα κάνει η Κομισιόν. Ορισμός των ευπαθών καταναλωτών. Δηλαδή, ήδη είμαστε σε ένα πιο ευρύ φάσμα. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό τελειώνω με δύο-τρεις άλλους τομείς που εμένα με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Πρώτον, η εφαρμογή. Σε εθνικό επίπεδο οι εθνικοί ρυθμιστές έχουν περισσότερες εξουσίες και πρέπει να έχουν τους πόρους και τη βάση για να λειτουργούν σωστά σε εφαρμογή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η υπηρεσία δεν έχει πολλές εξουσίες. Ωστόσο, έχει σε ορισμένες περιπτώσεις και μπορεί να επηρεάσει και να πείσει. Η συνεργασία με την Κομισιόν αποδεικνύει ότι μπορεί να οριστούν κανόνες και αυτό θα βοηθήσει. Δεύτερο, διαβούλευση. Από εμπειρία ξέρω ότι η προσπάθεια, ενδιαφερόμενη όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δίνουν τη γνώμη τους είναι σημαντικό. Αυτό που ήδη αποφασίσαμε το μεταφράσαμε σε περισσότερες διαδικασίες φιλικές όσον αφορά τη διαβούλευση για τους 500 εκατομμύρια αγορά καταναλωτών έτσι ώστε να έχουμε λογικές ρυθμίσεις. Τρίτον, υπάρχουν άλλα θέματα. Ο Γενικός Διευθυντής για την έρευνα όσο τον άκουσα τουλάχιστον σήμερα, από κομψότητα δεν ανάφερε κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Smart grips. Τι σημαίνει αυτό. Πολλές λέξεις για τις οποίες πολλοί νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά δεν ξέρουν. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν τεράστιες επενδύσεις στην Ευρώπη, σε συγκεκριμένα επίπεδα, ιδιαίτερα αφορά την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια στον εφοδιασμό, τα έξυπνα δίκτυα, smart grids, τα έξυπνα δίκτυα είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική λέξη και έννοια. Και τέλος, η Ευρώπη είναι περίεργο αλλά δεν είναι νησί. Δηλαδή η Ευρώπη πρέπει να κοιτάξει και προς τα έξω. Και τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιούμε ως ρυθμιστές ότι αυτό που ήταν στο παρελθόν κλειστό σύστημα όσον αφορά το αέριο και τον ηλεκτρισμό. Αυτό έχει αλλάξει. Και με ανανεώσιμε μορφέ ενέργειας και πάλι παρόλα αυτά θα εξαρτώμεθα από τους γείτονές μας για εφοδιασμό. Έπειτα, τα προβλήματα αυτά δεν είναι μόνο ευρωπαϊκά. Το LNG, ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο κλπ. Αφορούν και άλλους, άρα πρέπει να δούμε πέραν της Ευρώπης. και λίγο διαφήμιση. Στις 19 Οκτωβρίου στην Αθήνα έχουμε το Παγκόσμιο Φόρουμ Ρυθμιστών της Ενέργειας. Περίπου χίλια άνθρωποι θα είναι εκεί στην Αθήνα για να συζητήσουν ένα σωρό θέματα, από όπου ελπίζουμε τα στοιχεία να μας διευρύνουν τους ορίζοντες όσον αφορά τις διεθνείς θέσεις. Συνεργασία λοιπόν και συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Μεσόγειο, με την Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Ρωσία. Σε πολλούς τομείς δηλαδή κοιτάμε πέρα από τα σύνορά μας. Και προτιμά εδώ κύριε Πρόεδρε να σταματήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά για την υπενθύμηση των όσων κάναμε και τον όσο μας περιμένουν στους προσεχείς μήνες. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα έχετε εσείς την ευκαιρία να υποβάλλετε ερωτήσει, παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Εκεί πίσω ο πρώτος ομιλητής, μόνο που δυστυχώς δεν μπορώ να πω το όνομά σας. Κύριε Σλίτερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα θέλω να σημειώσω ότι συνεργαζόμαστε και με τους ε, προμηθευτές ε, των ε, μέσων αλλά και με τους καταναλωτές. Από τη μια λοιπόν υπάρχει από την πλευρά του προμηθευτή σαφής παρουσία, αλλά το κοινό δεν έχει έλεγχο των ρυθμιστικών σωμάτων, δεν έχει σαφή παρουσία στα ρυθμιστικά σώματα. Πώς λοιπόν θα μπορούσε το κοινό να συμβάλλει, να συμμετάσχει στη ρύθμιση των μέσων μας και Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Μόγκ, αφού δεν βλέπω κανένας άλλος να ζητάει το λόγο και αφού είναι μια ερώτηση μάλλον εκτεταμένης ε, εμβέλειας, ίσως θα ήταν καλό να απαντήσετε αμέσως. Ο κύριος Μόγκ, ε, άκουσα τον, τον όρο μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι το θέμα αυτό, με την, ενέργεια, με την ενέργεια και φαντάζομαι για την ενέργεια θα θέλετε να ρωτήσετε. Να απαντήσω λοιπόν ως εξής. Καταρχάς η ενέργεια είναι Περίπλοκο τομέα. δύσκολο να εξηγηθεί δηλαδή στον μη εμπειρογνώμονα και σα ομολογώ ότι εγώ ω μη εμπειρογνώμων βλέπω ότι είναι όντως μεγάλη πρόκληση. Έχουμε ένα πολύ καλό, εύχριστο ε, στο χώρο που ενθαρρύνει τον χρήστη να το χρησιμοποιήσει. Αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κανείς απόλυτα στη να το κάνει. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, ε, προσπαθούμε να διευκολύνουμε φυσικά στη διαδικασία την συμμετοχή και του κοινού και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι να αναπτύξουμε το σύστημα των, της επικοινωνίας ε, της ε, μετάδοσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να διευκολύνουμε και την παρουσία, τη συμμετοχή του κοινού. Τώρα έχουμε το δεύτερο τέτοιο ευρύ φόρουμ, έτσι ώστε να έχουμε τον καταναλωτή παρόντα ε, και να ακούσουμε τη γνώμη του. Τρίτον, έχουμε και νέα τεχνολογία στη θέσή μας και πάλι για να μιλήσω από τη σκοπιά της δικής μου Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής. Έχουμε διάφορες ομάδες ε, καταναλωτών σε πάνελ και πραγματογνώμονες σε διάφορες τις ομάδες εργασίας που ε, βοηθούν στην κατανόηση των περίπλοκων ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε. Και η δική μου δουλειά και εδώ στις Βρυξέλλες είναι να εξετάζουμε πολύ περίπλοκα τεχνικά ζητήματα και συνήθως το επιχείρημα προβάλλεται είναι «Α, δεν μπορεί ο κοινό θνητός να το καταλάβει». Όχι, δεν συμφωνώ εγώ με το επιχείρημα αυτό διότι θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη των ίδιων των ρυθμιστικών αρχών, των ίδιων των παραγόντων στον τομέα της ενέργειας, να εξηγήσουν, να βοηθήσουν τον κοινό θνητό να καταλάβει την κατάσταση. Και εν τέλει, η διαβούλευση για συγκεκριμένες ε, προσεγγίσεις ή τομείς της πολιτικής έχει μεγάλη σημασία. Ένα παράδειγμα, ο λογαριασμός. Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με το λογαριασμό σας του ηλεκτρικού, και τα λοιπά, τις ενέργειες δηλαδή, ε, και θέλετε να αμφισβητήσετε κάποιο κεφάλαιο, κάποιο σημείο του ε, λογαριασμού. Ειδικά δε όταν έχουμε προβλήματα και οικονομικά, δυσκολίες δηλαδή μερικές φορές λόγω των υψηλών λογαριασμών να τους ε, πληρώσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η κατάλληλη, το κατάλληλο σημείο επαφής με επαρκή χρόνο, με επαρκή εξηγήσει, αλλά ασφαλώς, για να βάλω και το χέρι στην καρδιά, Πολλά ακόμα έχουμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμψον, παρακαλώ. Η κυρία Τόμψον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση πολύ σύντομα. Είπατε ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές αντελήφθησαν, συμφώνησαν ότι εξαρτώμεθα από τους γείτονές μας για την προμηθή που προσπαθείτε ως σώμα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών να ξεπεράσετε τα στενά όρια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ακριβώς τι εννοείτε με τα λόγια αυτά και αν εννοείτε και την ε, συμφωνία για την ενέργεια στον ανατολικό χώρο της Ευρώπης. Ευχαριστώ κυρία Τόμψον που απαντήσατε εν μέρη στην ερώτησή σας. Ασφαλώς και έχει σχέση με, την, ε, ε, με τις ε, ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ενέργεια, αλλά εν μέρη μόνο. Καταρχάς προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας. Η προμήθεια σε ενέργεια και η ασφάλεια της προμήθειας είναι μεγάλο ζήτημα, και ιδιαίτερα όταν βγαίνουμε από τα σύνορα της Ευρώπης. Η ανανεώσιμες πηγές, η παραγωγή και η διανομή γίνονται όλο και περισσότερο πτυχή ή καθημερινή πτυχή και χαρακτηριστικό της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρώπης. Ένα από τα αισθήματα λοιπόν που με ε, ενδιαφέρουν είναι να ε, φροντίσουμε αυτές οι ανανεώσιμες πηγές να μπουν στην ε, Ευρώπη. Μεγάλη πρόκληση για μας, για το περιβάλλον, για την Ευρώπη την ίδια. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διευρύνουμε το δίκτυο της διανομής. Δεύτερον, η Ευρώπη είναι αδιαφανής. Παράδειγμα, εγώ ήρθα στους ρυθμιστές πριν από 6,5 χρόνια και στον πρώτο χειμώνα είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού και αφελώς ρώτησα τι γίνεται στην υπηρετική Ευρώπη για στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς έπρεπε να στηριχτούμε σε άρθρα από εφημερίδες, ελάχιστες δηλαδή πληροφορίες για το ποια ήταν η κατάσταση στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ και θα αλλάξει κι άλλο. Τώρα θα έχουμε διαφάνεια με την αναθεώρηση, στρατηγική αναθεώρηση της Κομισιόν και θα ξέρουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ενοποιημένο σύστημα, ένα ενιαίο σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μια καλή βάση στην Ευρώπη να μην εξαρτώμεθα από το εξωτερικό. Η διαμάχη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πριν από δύο χρόνια. Δεν υπάρχουν ακόμη και σήμερα ανησυχίε και αβεβαιότητα. Αυτό δείχνει ότι εξαρτώμεθα πάρα πολύ από το διάλογο μεταξύ Κομισιόν και Ρωσίας να ξέρουμε τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει ή να μην κάνει η ΓΚΑΣΠΡΟΜ. Η Κομισιόν βέβαια θα τα αποφασίσει αυτά. Υπάρχει μια ομάδα συντονισμού για το αέριο που επιτρέπει αξιολόγηση των δυσκολιών. Και πολλά μέτρα από εκεί θα βοηθήσουν. Πάμε χάρη στο παρελθόν το αέριο πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση στον αγωγό. Μερικές χώρες κατάφεραν να αντιστρέψουν τη ροή για να βοηθηθούν χώρες που έχουν προβλήματα, Ιταλία, Αυστρία. Πρέπει να δούμε πέρα από το ρωσικό εφοδιασμό. Έχουμε το νορβηγικό εφοδιασμό. Η Νορβηγία είναι μέτρος όχι ρυθμιστής, αλλά είναι μέλος του ΣΥΑ και του ΕΡΓΕΚ ως παρατηρητής και βόηθησε πάρα πολύ στις συζητήσεις μας όσον αφορά τα αριθμιστικά θέματα. Επιπλέον, από εκεί και πέρα μάλλον, αφορά τις, τα κράτη-μέλη και, και την Κομισιόν. Εμείς ως ρυθμιστές φροντίζουμε η πληροφορία να είναι προσβάσιμη, κατανοητή και με συνεργασία να γίνονται όλα. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σνάφος Οντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για όλες αυτές τις εξηγήσει Πάρα πολύ ενδιαφέρουσε ήταν. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τα δίκτυα, ιδιαίτερα στον ηλεκτρισμό. Εμείς λέμε να ξεχωρίσουμε τα δίκτυα των παραγωγών και των διανομέων ενέργειας. Και στην Ένωση έχουμε δίκτυα που είναι ιδιοκτησία διαφόρων. Τι λέτε, πώς πρέπει να εφαρμόζει η νόμοι της αγοράς στα δίκτυα αυτά. Θα μας συνέφερε ως Ένωση πολιτικά τα δίκτυα αυτά, τα ηλεκτρικά δίκτυα, να ανήκουν σε μια δημόσια ευρωπαϊκή αρχή, έτσι ώστε οι πολίτες να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα δίκτυα δεν θα πέσουν στα χέρια μιας, ε, ενός καπιταλιστή ιδιοκτήτη όπως η Gazprom ή κάποιος άλλος. Ποια είναι η άποψή σας για την παραγωγή, άσχετα με τη διανομή. Αυτόν τη συμπεριφορά την παρακολουθείτε. Δεύτερη ερώτηση για το αέριο. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν να γίνει μια εταιρεία αγοράς αερίου από τον Κάφκασο. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Και αν η πρόταση αυτή, υπάρχει πρόταση χώρας μέλους να γίνει μια, ένας ευρωπαϊκός κεντρικός σταθμός αγοράς αερίου για να βαρύνει στην τιμή του αερίου και να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό με την καλύτερη τιμή. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Απάντηση. Καταρχάς συγχαρητήρια για τις πολύ συγκεκριμένες σας ερωτήσεις. για την πρώτη. Νομίζω ότι γύρω από το τρίτο πακέτο ξεκίνησαν πολλές συζητήσεις και ζητήματα ως προς την αποδέσμευση και την διαμόρφωση του τομέα τόσο της ηλεκτρικής ε, ενέργειας και του φυσικού αερίου. και εν προκειμένου αναγνωρίστηκε ότι αρκετές φορές η ρυθμιστική διαδικασία αντικατοπτρίζει την κατάσταση του κάθε κράτους μέλους. Έτσι λοιπόν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ε, είδαμε τα θέματα λίγο πολύ όπως προκαλούσαν το ενδιαφέρον της πολιτικής ή της κοινή γνώμη. Θα δείτε ότι είναι ούτως ή άλλως θέματα σε μεγάλο βαθμό των κρατών μελών, αλλά βέβαια και του Κοινοβουλίου. Το να υπάρχει λοιπόν ένα ευρωπαϊκό σώμα το οποίο θα μπορούσε να τα απορροφήσει όλα αυτά, η πρότασή σας δηλαδή, σημαίνει ότι θα είχε κερδίσει και την εμπιστοσύνη των αγορών, το εν λόγω σώμα και των κυβερνήσεων, έτσι ώστε να, να λάβει την ε, επένδυση που χρειάζεται για την ενοποίηση, ενσωμάτωση, ολοκλήρωση των ε, αγορών ενέργειας στην Ευρώπη στοιχεία έχω να παρουσιάσω, όλες δεν είναι η στιγμή τώρα για τη δική μου τουλάχιστον αρχή, σε δύο εβδομάδες περίπου θα παρουσιάσω τα δικά της στοιχεία. Αλλά θα σας δώσω κάποια στοιχεία από τους Ernst Young, την εταιρεία consulting. 30 δις στο Ηνωμένο Βασίλειο για την προσεχή δεκαετία χρειάζονται σε επενδύσεις. Έτσι, αν κάνει κανείς τη σχετική προβολή, σε αναλογία και των λοιπών δικτύων των άλλων κρατών μελών, είναι τεράστια. οι ανάγκε είναι τεράστιε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δύο ή τρία χρόνια είχε μιλήσει νομίζω για τρία-τρει. Τεράστια ποσά. Και δεν νομίζω ότι είναι ε, ευχερέ το να εξασφαλιστούν τα κονδύλια αυτά, ούτε σε κρατών μελών ασφαλών, αλλά ούτε και κοινοβούλιο πίσω τα στήσει λεφτά αυτά από τον Ευρωπαίο πολίτη, από το φορολογούμενο. Επίσης για το τρίτο αυτό πακέτο βλέπουμε τα πλεονεκτήματα μιας απελευθερωμένης αγοράς. Εγώ έχω δράσει, έχω αρκετά χρόνια πίσω μου σε μια απελευθερωμένη αγορά, αλλά θα ήθελα να σημειώσω ότι υπάρχουν κάποια σημεία, με όλα τα καλά που έχει η απελευθερωμένη αγορά, όπου χρειάζεται παρέμβαση, ρύθμιση και για την ασφάλεια των προμηθειών ασφαλώς και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και άλλες αγορές ε, και, και σε άλλους τομείς. Επίσης, ο κίνδυνος της Gazprom, βέβαια ίσως να με διαψεύσει η ιστορία, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναβρυχηθεί η ρωσική αρκούδα και ότι ως εκ θα μπορέσουμε να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία και ένα πιο θετικό μέλλον στο θέμα αυτό. αλλά πάντως υπάρχουν ανησυχίες και ως προς τις επενδύσεις και ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων από πλευράς Ευρώπης, γιατί η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Η Γαλλία, παραδείγματι, έχει διαφορετικές συνθήκες από πολλά άλλα κράτη-μέλη, αφού έχει τόσο μεγάλο ποσοστό παραγωγής ενέργειας από, το, τα πυρηνικά. Και μάλιστα την εξάγει και όλα σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και δική μου. Έτσι λοιπόν, η Ευρώπη με την προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς, με την ανάπτυξη των διασυνδέσεων, με τις ανανεώσιμες πηγές, την αιωλική ενέργεια, στην ε, Βόρεια Θάλασσα ιδιαίτερα που καλύπτει αρκετές χώρες, εξασφαλίσει περισσότερη ασφάλεια. Αντίστοιχα αναφερθήκατε και στο φυσικό αέριο. Είχαμε μάλιστα εμείς μία... Έχουμε μάλλον τη Γενική Συνέλευση αύριο των ρυθμιστικών αρχών με θέμα στην ημερήσια διάταξη ακριβώς στην διατύπωση των απόψεών μας και προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα σώμα κεντρικό το οποίο θα αναλαμβάνει την αγορά αερίου. Αλλά προς το παρόν δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο. Εάν χρειαστεί να μελετήσουμε περισσότερο την υπόθεση, ίσως ο βαθμός συνεργασίας να είναι μάλλον αδύνατο, γιατί όταν κανείς έχει τόσο τόση ιστορία, τόση εμπειρία στην υπόθεση αυτή όπως εγώ, ίσως είναι πολύ πιο δύσπιστος ή λιγότερο αισιόδοξο. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, ώστε να μην καταφέρουμε και ποτέ να φτάσουμε στον απόλυτο βαθμό συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο για τις εξηγήσεις και υποφελούμε της ευκαιρίας που είστε εδώ και θα σα κάνω μια ερώτηση που αφορά τη χώρα μου. Μια απέτηση εκ μέρους ενός Γάλλου φορέα για να τη συνδέσει για επενδύσεις, επενδύσεις αναφέρθηκε σε λύσεις που ανακοινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, αν ζητείτε, ας πούμε, το 80% για το αέριο, 80% από βορρά προς νότο και τι ποσοστό για την κίνηση αντίστροφα. Πώς θα γίνει η σύνδεση αυτή. Αυτός ο όρος για μας μας εκπλήσει. Και δείχνει ότι πάνε να προστατευτεί μια εθνική αγορά. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. και τι θα γίνει, τι θα πιστεύετε ότι θα γίνει στο μέλλον σε παρόμοιες περιπτώσεις. Απάντηση. Ευχαριστώ κυρία Βιέρα Μαντουρέλ. Διότι η ερώτησή σας με επιτρέπει κάτι που θα έπρεπε να είχα πει στην εισαγωγή. Η Ευρώπη ως ενιαία αγορά και για την ενέργεια θα πρέπει να κάνει ένα βήμα μπρο σε σχέση με τη σημερινή κατακαιρματισμένη αγορά. Το Κοινοβούλιο, όταν ξεκίνησαν οι περιφερειακέ πρωτοβουλίε. ανησύχησε και σωστά, διότι υπάρχει αμφιβολία. Αντί να πάμε προς μία ενιαία αγορά, να έχουμε περιφερειακές αγορές. Άρα να συνεχίσει ο κατακαιρμένος κατακαιρματισμένος χαρακτήρας της ενεργειακής αγοράς. Ε, λοιπόν, εμείς πριν από μερικά χρόνια, πριν από μερικά χρόνια, ως ρυθμιστές επαναλαμβάνω, θελήσαμε να κινηθούμε προς το ενιαίο αυτό, προς το βήμα αυτό, προς την ενιαία αγορά, είναι τεράστιο βήμα και έπρεπε να πείσουμε την Κομισιόν. Γι' αυτό πήραμε περιφερειακές πρωτοβουλίες. Αυτό ξέχασα να πω στην εισαγωγή μου. Αυτό επέτρεψε περιφέρειες με ανάλογο βαθμό επιτυχίας. Αλλού είχαμε ε, ε, συμμετοχή των κυβερνήσεων, αλλά όχι, να σημειώσουν πρόοδο σε συνεργασία στην περιφέρεια αυτή. Αυτό βοηθάει στον εφοδιασμό σε ενέργεια, σε αποδοτική χρήση της ενέργειας, γιατί η βόρεια αγορά, χάρη, είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, άρα μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο της. Επίσης κάτι άλλο, μια άλλη διαφήμιση. Έχουμε μια διάσκεψη για τις περιφερειακές πρωτοβουλίες. Κάποιος βουλευτής δικός σας θα είναι παρόν από ό,τι ξέρω και θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Αφορά ιδιαίτερα την Ιβυρική Χερσόνησο, την Νότια Ευρώπη. Βέβαια, ακόμα ως ομάδα δεν το συζητήσαμε. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να δουν τι μπορεί να γίνει παραπάνω στις περιφέρειες. Η συγκεκριμένη ερώτηση. Υπάρχει ένας νέος κανονισμός, σχέδιο μάλλον κανονισμό της Κομισιόν για τον ασφαλή εφοδιασμό εμείς έχουμε επιφυλάξεις. Υπάρχουν μερικές όμως καλές αρχές όσον αφορά τη διαφάνεια, τη συνεργασία. Το κατά πόσο θα παρέμβει η Κομισιόν στη διαδικασία κλπ. Αυτό θα βοηθήσει σε σχέση με τις ακραίες περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε. Έπειτα θα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσον η υποδομή, ποια θα είναι η υποδομή που χρειάζεται και αν επαρκεί. Αν δούμε τις προδιαγραφές παροχής εφοδιασμού, θα πρέπει να εμείς ως ρυθμιστές θέλουμε αυτό να γίνει με βάση αξιολόγηση των κινδύνων. Να μην δοθούν χωρίς λόγο κονδύλια. Οι παρατηρήσεις σας δεν ξέρω αν αφορούν ειδικά τις σχέσεις Γαλλίας-Ισπανίας. Για πολλά χρόνια υπάρχουν δυσκολίες στη σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Ο καθηγητής Μόντι, ο πρώην Επίτροπος, πρόσφερε χρήσιμο έργο προκειμένου οι δύο πλευρές να συζητήσουν. Από τη μία μεριά, από τη Γαλλία, είχαμε τις ανησυχίες για επενδύσεις και μείωση των ποσών ενέργειας που έπρεπε να δώσει στην Ιβηρική. Από την ισπανική πλευρά ο προβληματισμός ήταν να υπάρχει επαρκής εφοδιασμός. Εμείς, μάλλον ως Ευρωπαίος συντονιστής, ο καθηγητής Μόντι βόηθησε να λυθεί αυτό το περίπλοκο πρόβλημα. Ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες, τις προσθέτες ε, εξηγήσεις, επίσης και τους συναδέλφους και τις ερωτήσεις τους. Υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να υποβάλει μια ερώτηση, χρειάζεται κάποια διευκρίνηση. Εάν όχι, μπορούμε νομίζω να κλείσουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Να ευχαριστώ τον κύριο Μόκ, τον Λόρδο Μόρκ, για την παρουσία του, τον χρόνο που μας διέθεσε και τις πληροφορίες που μας έδωσε. Και ασφαλώς κατά τη διάρκεια της θητείας θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να συνασμιλθούμε. Τα θέματα έχουν δυστυχώς ακόμη πολλά κοινά δεν έχουν αριθμιστεί ακόμη. Σας ευχαριστώ πολύ και έτσι κηρύσω το θέμα, την ε, λήξη της συνεδριάσεως μας. Για να ε, ξεκινήσουμε το ταχύτερο δυνατό τους, ε, τη συνεδρία των συντονιστών.